say that this is yeah, one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, ακρόασης για τις νέες ε, για τους νέους κανονισμούς σε δημοσιονομικό επίπεδο απολογισμός και για χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μάλλον, απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις. λοιπόν, πρόκειται για τον απολογισμό μιας ε, έντονης και εργόδους σειράς νομοθετημάτων στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πολλές ε, πράξεις έχουν εγκριθεί στα τελευταία χρόνια και πρέπει να τις εξετάσουμε και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα και την αλληλοδιαπλοκή τους και επίσης πρέπει να δούμε τις ε, μελλοντικέ προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη βάση αυτού του απολογισμού και φυσικά είναι το CMU που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί και νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ένωση των ε, για τις κεφαλαίες αγορές. Πιστεύω ότι τώρα η Κομισιόν έχει τη θέληση να μας δώσει αυτό τον απολογισμό, αυτή την αξιολόγηση και η πρωτοβουλία της θα πρέπει να συνδέεται με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες. Είναι χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρχίσει να εργάζεται για το θέμα αυτό και ένας καλός τρόπος να ξεκινήσουμε είναι με το να αναλύσουμε το θέμα σε βάθος. Και είναι πολύ χρήσιμο που ο εισηγητής έτεινε να διενεργηθεί αυτή η δημόσια κρόαση. Έχουμε πολύ καλούς εμπειρογνώμενους εδώ. Ξεκινάμε δίνοντας το λόγο στους τέσσερις ομιλητές για τέσσερα λεπτά στον καθένα και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. ξεκινάμε με τον Μάρτιν Γκρουλ ο οποίος είναι ο, ο υπεύθυνος του χρηματοπιστωτικού τμήματος της Raiffeisen International. Έχετε το λόγο κύριε Γκρούλ. Γκρούλ, έντιμα, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες για την πρόσκλησή σας να έρθω σε αυτή την ακρόαση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Λέγομαι Μάρτιν Γκριλ και είμαι ο επικεφαλής του λογιστικού τμήματος της Raiffeisen Bank International που έχουμε έδρα στη Βιέννη και η Κεντροανατολική Ευρώπη είναι η κύρια αγορά μας. Για περίπου 25 χρόνια η Raiffeisen International λειτουργεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε 17 αγορές με 54.000 εργαζομένους και καλύπτουμε περίπου 15 εκατομμύρια πελάτες. Από την οπτική γωνία μιας φυσιολογικής εμπορικής τράπεζας, νομίζω ότι το θέμα της ακροασής σας είναι πάρα πολύ σωστό για μας. Ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση θα δώσει μια βάση στην υγεία του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα, ο οποίο είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο για μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Είναι απαραίτητο όμω αυτό το ρυθμιστικό περιβάλλον να μην, συνθλίπει, να μην συνθλίψει τις ε, τράπεζες και εταιρείε στον τομέα αυτό και να τις εμποδίσει να δρουν αποτελεσματικά. Ας συνοψίσω τα κύρια προβλήματα, τα κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος αν θέλετε που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τράπεζες. Χαμηλά επιτόκια, μικρή ε, ζήτηση για πιστοδοσία και προϋπολογισμοί που είναι απρόβλεπτοι, χαμηλή κερδοφορία και περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων, όλο και περισσότερες απαιτήσει για κεφαλογική επάρκεια και επίσης πρόσθετες ε, ε, εισφορές και τέλη που εισάγονται στα πλαίσια της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Με ένα τέτοιο πλαίσιο έχουμε κέρδιες προκλήσεις για όλο τον οικονομικό αυτό τομέα που μπορούν σε τελική ανάλυση να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη. Οι απαιτήσει σε κεφαλουχικό και επίπεδο ρευστότητα τη CRD4 και CRR και η Τραπεζική Ένωση είναι σημαντικά βήματα για να μπορέσει να ενισχυθεί η σταθερότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Στο μέλλον δεν πρέπει οι φορολογούμενοι να επομίζονται το βάρο τη ανάκαμψη και τη επίλυση μια τράπεζα. Αλλά προπόθεση για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα στην πράξη είναι μια σωστή περίοδο εφαρμογή για να δημιουργηθεί το απαραίτητο κεφάλαιο μετοχικού χαρακτήρα. Αλλιώ η δανειοδότηση τη οικονομία θα μειωθεί και αυτό θα παραλύσει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι σαφέ ότι οι επόπτε έχουν την τάση να επιταχύνουν την εφαρμογή αυτών των μέτρων και ζητούν αποθεμάτα σε επίπεδο κεφαλαίου πολύ πιο νωρί από ό,τι απαιτεί η νομοθεσία. Οι τελευταίε εξελίξει σε σχέση με τη Βασιλεία 4 μπορεί ακόμα και να ενισχύσουν αυτή την τάση και να εμποδίσουν ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση των πελατών μας. Οι νέες προτάσεις αυξάνουν τη στάθμιση του κινδύνου και αυτό περιορίζει την ε, δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ακόμα περισσότερο. Ας μην ξεχάσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να αναφέρω επίση τρει τομεί όπου υπάρχει έλλειψη συνεκτικότητας του τωρινού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου που έχουν σαν ε, αποτέλεσμα την τροχοπέδηση της χρήσης ανθρωπίνου και οικονομικού κεφαλαίου και κάνουν πιο δύσκολο για τις, για τις τράπεζες να δανειοδοτούν. Πρώτα απ' όλα, οι υποχρεώσεις παροχής αναφορών. Τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για την παροχή αναφορών καλύπτουν περίπου 1.800 σελίδες. Υπάρχουν διάφορες αρχές, η Κεντρική Τράπεζα, οι Εθνικές Αρχές, ο Φορέας ε, επίλυσης και ανάκαμψης, ο ενιαίος που θα πρέπει να συντονίσουν τις διάφορες δραστηριότητες. Όπως έχουμε τονίσει στο παρελθόν, μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση απαιτεί και σωστό συντονισμό μεταξύ των εφοπτικών αρχών. Σήμερα έχουμε μια επικάλυψη των <clears throat> αναγκών για παροχή αναφορών και επιπλέον στο άμεσο μέλλον θα αυξηθούν οι αιτήσει για παροχή αναφορών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να υπάρχουν αναφορέ για οποιοδήποτε δάνειο το οποίο ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ. Είναι φανερό ότι ιδίω οι μικρότερες τράπεζες θα έχουν τεράστιο άχθο με αυτές τις νέε απαιτήσει. Δεύτερο θέμα είναι οι απαιτήσει σε επίπεδο κεφαλαίου. Είναι σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση των απαιτήσεων κεφαλογικής επάρκειας σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί παραμένει ακόμα υψηλός βαθμός αβεβαιότητας. Παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα σαφές πώς ενσωματώνονται οι εθνικές απαιτήσει για κεφαλογική επάρκεια στο πλαίσιο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει ένα σαφέ και συνεκτικό πλαίσιο για να καθορίζονται και να εφαρμόζονται οι, τα περιθώρια κεφαλογική επάρκεια. Για τι μικρότερε τράπεζε είναι απαραίτητο οι υποπτικέ αρχέ να προσαρμόσουν τι ρυθμιστικέ ανάγκε στο επιχειρηματικό τη μοντέλο. Μια μικρότερη τράπεζα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να υπόκειται στι ίδιε αιτήσει που ισχύουν για τι μεγαλύτερε τράπεζε, παραδείγματο χάρη παροχή αναφορών, εσωτερική διακυβέρνηση και πολιτικέ ε, αμοιβή των στελεχών. Ένα δεύτερο θέμα <clears throat> και σας ζητώ συγγνώμη γιατί ίσως θα ξεπεράσω τα πέντε λεπτά. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα αλλά και πολύ σημαντικό. Τα τέλη που επιβάλλονται στις τράπεζες μειώνουν τη σταθερότητα και φέρνουν ένα αμφιβόλο την ενία αγορά και την, ε, τον ισοδίκαιο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη αύξηση στα τέλη που επιβάλλονται στις εθνικές τράπεζες με το στόχο να μην είναι οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν για την κατάρρευση των τραπεζών. Υπάρχει φορολογία αυτή τη στιγμή των τραπεζών σε εθνικό επίπεδο σε 16 χώρες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο για τα τραπεζικά τέλη και δημιουργεί πολλά προβλήματα στις διαμεθοριακά λειτουργούσες τράπεζες. Στο Ρωμένο Βασίλειο Παγμοσχάρη, ορισμένα τέλη είναι φόροι που χρηματοδοτούν το γενικό προϋπολογισμό. Στη Γερμανία είναι ε, τέλη τα οποία τροφοδοτούν ένα ε, ταμείο επίλυσης των τραπεζών που είναι χωριστός από τον προϋπολογισμό. Πολλοί από αυτού τους φόρους πληρώνονται επί τη βάση των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας ανεξάρτητα από την κερδοφορία μιας τράπεζας. Και επίσης είναι πρόβλημα ότι κάποιοι από αυτούς τους φόρους πληρώνονται επιπλέον των συνεισφορών στον εθνικό ή στο ευρωπαϊκό το ευρωπαϊκό ταμείο επίλυσης και ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα αβάστακτο βάρος γιατί τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να αυξάνουν την κεφαλουχική μας βάση για περισσότερη δανειοδότηση και για νέα μοντέλα εξυπηρέτησης των πελατών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει ο εθνικός φόρος της τράπεζας να χρησιμοποιείται σαν συνεισφορά στο Ταμείο Επίλυσης, Ευρωπαϊκό και Εθνικό και στο μέλλον θα πρέπει αυτό να είναι το μόνο εργαλείο το Ταμείο αυτό για να εξασφαλίσει τα των χρηματοπιστωτικών αγορών και να σπάσει τη σύνδεση μεταξύ κρατικού χρέους φορολογουμένων και ε, κατάρρευσης τραπεζών. Για μια ομάδα διαμεθοριακών δραστηριοτήτων όπως εμείς <clears throat> που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζώνη ευρώ και μη ζώνη ευρώ είναι απαραίτητο να υπάρξει εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών για ένα λειτουργικό επιχειρηματικό μοντέλο. Την πράξη όμως είναι πολύ διαφορετικές αυτές οι πρακτικές από χώρα σε χώρα όπως πολύ σωστά το έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην έκθεσή της του Απριλίου 2015. Οι αποφάσεις σε σχέση με τα ΣΡΕΠ, δηλαδή τις ειδικέ εποπτικές ανάγκες που απορρέουν από, από την οδηγία CRD4. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που έχουν οι τράπεζες και σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις ζητούν ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίου λαμβάνοντα υπόψη το προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο καθορίζεται αυτό το ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίου και εφαρμόζεται σε φορεί είναι πολύ διαφορετικό. Μερικέ αρχέ προτιμούν να το αναφέρουν με τη μορφή μια προσδοκία ή μια σύσταση, άλλε θεωρούν ότι αυτό το ελάχιστο επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστεί ω νομικά δεσμευτική υποχρέωση αυτή η έλλειψη ομοιογένεια στην λήψη απόφαση οδηγεί σε ανισότητα ανταγωνισμού και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Οι πρακτικέ εποπτεία επίση είναι διαφορετικέ σε ό,τι αφορά την ε, διαθεσιμότητα κεφαλιακών εργαλείων που μπορούν να επιτυχούν του επιδιωκόμενους στόχου. Ορισμένε αρχέ είναι περιοριστικέ, άλλε είναι πιο χαλαρέ σε σχέση με το φάσμα των εργαλείων. Τέλο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στι νέε αλλαγές που έχουν γίνει με το σύστημα IFRS, το νέο σύστημα λογιστικής απεικόνησης. Το IFRS 9 συγκεκριμένα, το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα για τα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών. Λέουν ορισμένοι ε, αναλυτές ότι μπορεί να αυξήσει κατά 10 με 13% το απαιτούμενο κεφάλαιο στην τραπεζικό τομέα της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για όλα αυτά τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία μπορεί να εγκριθούν στους επόμενους μήνες. Και έρχομαι στο τέλος και πάλι σας ζητώ συγγνώμη για την μακρηγορία μου. Θέλω να τονίσω ότι χρειάζονται μια ανάσα οι τράπεζε. Θα πρέπει να του δοθεί αρκετό χρόνο για αξιολόγηση του, των τωρινών κανονισμών για τη χρηματοπιστωτική αγορά και για καλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση. <clears throat> θα πρέπει να, τα εθνικά τέλη τη τράπεζα να πηγαίνουν στο Ταμείο Επίλυση και Ανάκαμψη. Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται κάτι περισσότερο από χρηματοπιστωτική σταθερότητα και καλύτερη ρύθμιση. Χρειάζεται οι τράπεζε να έχουν έσοδα για να μπορούν να παίξουν το ρόλο του ω χρηματοδοτική ενδιάμεση που θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Καέλα Κόλερ. Γενική Διευθύντρια από το Insurance Europe. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Πρόεδρε Παλτιέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που, καλήσα, καλέσατε και τον τομέα των ασφαλίσεων. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις και θα ήθελα να δείτε σας παρακαλώ και τα έγγραφα που δώσαμε στη γραμματεία, τα οποία ακριβώς βοηθάνε να καταλάβετε καλύτερα αυτά που θα σας πω. Από πλευράς λοιπόν ασφαλίσεων θέλω εδώ να υπογραμμίσω τρία θέματα κλειδί και τρει προκλήσεις. Πρώτον, μεγάλος φόρτο πληροφοριών και πώς χρησιμοποιούνται στις διαδικασίε επιλογής των προϊόντων. Δεύτερον, πώς θα δουλέψει το Solvency 2 και τρίτον, να ετοιμάσουμε διεθνεί προδιαγραφέ με ισχυρή ευρωπαϊκή εντολή. Έρχομαι στο πρώτο μου θέμα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον υπερβολικό φόρτο πληροφοριών και τις επικαλύψεις που λαμβάνουν χώρα πολλές φορές σε διάφορα νομοθετικά κείμενα. Ε, υπάρχουν λοιπόν ασφαλίσεις οι οποίες βασίζονται σε επενδυτικά προϊόντα. Υπάρχουν πέντε νομοθετικά κείμενα που προβλέπονται για το μέλλον. Το MD2, το ΣΥΣ, το Solvency 2, το Distance Marketing Directive και η οδηγία e-commerce. Η δουλειά έχει επικεντρωθεί βέβαια στα επιμέρους νομοθετικά κείμενα, αλλά υπάρχει και μια συνδυασμένη επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σήμερα έχουμε 74 απαιτήσει πριν από τη σύναψη αλλά 147 θα είναι αυτές στο μέλλον. Συνεπώς θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας κατά 183% έως και 330%. Και, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό εδώ, υπάρχουν ε, επικαλύψεις, απαιτήσει για επικαλύψεις δηλαδή, γιατί πολλά κείμενα περιλαμβάνουν τους ίδιους κανόνες, παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται για το IMD2. Έρχομαι τώρα στην οδηγία Solvency 2. Όπως ξέρετε, ο κλάδος στήριξε την ενημέρωση του πλαισίου Solvency με ένα πιο εξυγχρονισμένο σύστημα όπως είναι το Solvency 2. Η διαδικασία ήταν μακρά και περίπλοκη. Κράτησε 14 χρόνια περίπου. Τρεις είναι οι ανησυχίες μας. Πρώτον, βασίζεται σε μια αρχή το σύστημα αυτό, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 3.000 σελίδες Επεξηγήσει για τα εργαλεία. Δεύτερον, η αρχή τη αναλογικότητα δεν λειτουργεί όπω αρχικά ε, πρόκειται να λειτουργήσει και δεν αντικατοπτρίζονται οι πραγματικέ ανάγκες της αγοράς, κάτι το οποίο βέβαια επηρεάζει τι επενδύσει μακροπρόθεσμα και οδηγεί και σε μια μεταφορά των κινδύνων από τον κλάδο ε, στους ιδιώτες. Κάτι το οποίο βέβαια ισχύει για τους μελλοντικού συνταξιούχους. Άρα η πρόκληση είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα και στο 1 αλλά και στα 2 και 3 και πιστεύουμε ότι η ευκαιρία είναι να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την Κεφαλαϊκή Ένωση αλλά ελπίζουμε ότι τα θέματα τα οποία σας ανέφερα θα αντιμετωπιστούν μέχρι το 2018. Έρχομαι Τώρα, στο τρίτο ζήτημα, που είναι πώς θα ετοιμάσουμε διεθνείς προδιαγραφές με μια ισχυρή ευρωπαϊκή εντολή. Το 2013, η Διεθνής Ένωση Παροχών Ασφαλίσεων είχε μιλήσει για τρεις προδιαγραφές που θα αναπτυχθούν μέχρι το 2016, σε τρία χρόνια δηλαδή από τότε. Και αυτό σήμαινε ότι οι προδιαγραφές αυτές θα έπρεπε να αναπτυχθούν γρήγορα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόσετε δηλαδή το Solvency 2. Η ανησυχία είναι ότι το περιθώριο ελιγμών για τους νομοθέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι περιορισμένο γιατί οι προδιαγραφές αυτές ζητούν εφαρμογή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό θα οδηγούσε σε αλλαγές του Solvency 2 που θα επηρεάζανε όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Γι' αυτό από τη δικιά μας την πλευρά είναι πολύ βασικό οι διαπραγματευτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μιλούν μόνο με μία φωνή, αλλά οι διαπραγματεύσεις αυτές να γίνονται με διαφάνεια. Σήμερα, όσον αφορά εμάς, δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια εντολή. Και ποιο είναι το περιεχόμενό της. Κάποιες προδιαγραφές εγκρίνονται σε διεθνές επίπεδο, αλλά παραμένουν άλλες δύο προδιαγραφές που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και με την βοήθεια του σώματος αυτού για να αντιμετωπιστούν ακριβώς ε, οι δυσκολίες που παραμένουν. Τέλος, για την ΕΙΟΠΑ. Εμείς στηρίζουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχή για τις ε, ασφαλίσεις και τα ταξιδιωτικά και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν θέματα όπως είναι η διακυβέρνηση, η εποπτεία και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα επίπεδα θα στηρίξουν την εφαρμογή της πολιτικής που θα ληφθεί από του συνομοθέτες. Όλα αυτά τα ζητήματα όπως τα παρουσίασα μπορούν να αντιμετωπιστούν και ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δουλέψει προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε στον Νίαμ Μόλενεϊ, καθηγητή στο London School of Economics και αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Βουλίου κυρίες, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη, ε, με μεγάλη χαρά θα μιλήσω ενώπιον του Κοινοβουλίου σε αυτήν την ε, ε, κρίσιμη περίοδο. Ε, ίσως είναι ακόμα νωρίς έτσι ώστε να κάνουμε έναν γενικό απολογισμό ε, όσον αφορά την ε, κρίση γενικότερα. Ωστόσο ε, ήρθε η ώρα έτσι ώστε να κάνουμε έναν απολογισμό σχετικά με την δημιουργία της ε, κρίσης αυτής. νομίζω ότι το ρολόι πλέον χτυπάει αρνητικά όσον αφορά τους ελέγχους, κυρίως όσον αφορά τις κεφαλαίες αγορές. Απ' την άλλη πλευρά ε, η απέτηση ή μάλλον το, ο, ο, ο βαθμός ε, ρύθμισης ε, που απαιτείται όπως αποδεικνύεται από σειρά αποτυχιών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής μελέτης. Και κατά αυτή την έννοια η εργασία της ΕΚΟΝ είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, έχω τρία σημεία όσον αφορά την ρύθμιση των χρηματαγορών για τα επόμενα ε, και τις χρηματοπιστικές υπηρεσίες για τα επόμενα χρόνια από τη μία η εποπτεία και από την άλλη η ανάγκη να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να δούμε ε, γενικά ε, το οικοσύστημα, τον, το θεσμικό το οποίο είναι ευάλωτο. Η Τραπεζική Ένωση και ο ΙΕΦΣΕΦ έχουν δημιουργηθεί χωρίς να έχουν πάρα πολύ ισχυρές ε, ε, βάσεις. Ιδιαίτερος δε η EBA, η Αρχή Τραπεζικής Εποπτείας, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ε, την ενιαία αγορά. Οποιαδήποτε, ε, οποιαδήποτε παρέκκληση στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε άμεσα, ενδεχομένως και με άμεσες μεταρρυθμίσεις οπουδήποτε αυτό είναι απαραίτητο. Είναι πολλά τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν τη χειραγώγηση της αγοράς ε, και βεβαίως ε, η ε, προστασία των καταναλωτών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και κινδυνεύει να παραβλεφθεί εάν αναφερθούμε μονάχα στις ίδιες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τώρα το πραγματικό έργο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα ESAs που μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο και ιδίω όσον αφορά τις ε, ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις. Ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει ανεξάρτητη διακυβέρνηση η οποία θα παρακολουθείτε, όμως στενά. Τώρα θα μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε τα ESA να είναι πιο ευέλικτα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να δεχτούμε έναν συγκεκριμένο ας πούμε βαθμό ε, ε, επανάστασης αλλά με μικρό έψιλον ε, ε, που θα πρέπει να γίνει δηλαδή με ε, οργανωμένο, σχεδιασμένο και αναλογικό τρόπο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές περιπλοκές. Αντίστοιχα, η νέα σειρά ε, review clauses, ε, ρητρών αναθεώρησης, ε, είναι απαραίτητο να υπάρχουν. Η διαδικασία αναθεώρησης θα μπορούσε ας πούμε να ε, αντιμετωπίσει νομικά, νομοθετικά συγγνώμη, κυρίως ε, τις, ε, τους κινδύνους όσον αφορά τις επικαλύψεις και όσον αφορά τις ενδεχόμενες ανφιλεγόμενες απαιτήσει, καθώς επίσης και την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Θα μπορούσε επίσης να λάβει υπόψη τον ορισμό π.χ. του κεφαλαίου υπό το CRD4 ε, ή το καθεστώς CRR. Επίσης ε, η σαφήνεια ε, του περιμέτρου, της περιμέτρου εντός της οποίας ο ευρωπαϊκός κανονισμός θα λειτουργεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να συλλέγει ε, δεδομένα ε, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και άλλωστε αποτελεί και νομοθετική απέτηση σύμφωνα με τα νέα FINREP, COREP, τις απαιτήσει υπό το CRD4 και το CRR. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε καλύτερα τις ανάγκες πίεση και απαιτήσει των αγορών, αλλά χωρίς να λησμονούμε και τους ε, ε, ε, καταναλωτές και τους χρήστες. Το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω αφορά την προσέγγιση σε επιπλέον μεταρρυθμίσεις. Ο χρηματοπιστωτικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο όμως αποτελείται από πολλά ακόμα κινούμενα και όχι σταθεροποιημένα στοιχεία. Χρειάζεται βεβαίως νέος κανονισμός, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια των διαφόρων υπαρχουσών μορφών ε, ε, κανονισμού. Ε, θα πρέπει να προβλεφθούν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προχωρήσουν με ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Εν τέλει, ο Κρίστοφ Νίτζομ, Γενικός Γραμματέας του Finance Watch, θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάλτς, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που καλέσατε την Finance Watch να μοιραστεί μαζί σας κάποιες από τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών δομένες υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος ε, στο πλαίσιο τη εκτίμησης της γενικής κατάστασης ε, και των προκλήσεων που συνδέονται με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, να πω ότι κάποιες πιθανές μικρές επικαλύψεις είναι μικρό κόστος σε σχέση με τα ωφέλη σε σχέση με το κόστος της ανεπαρκούς νομοθετικής ρύθμισης. Η συνολική αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 θεώρησε ότι όλες οι επιμέρους νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες ήταν θετικές. Τρίτον, ε, αυτή η εκτίμηση της κατάστασης ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να οπισθοδρομήσουμε και να ελαφρύνουμε την νομοθεσία. Αντιθέτως, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα κενά και τις ασυνέπειες που υπάρχουν ε, στην ε, ε, χρηματοπιστωτική νομοθεσία για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας μετά την κρίση ήταν μικροπροληπτικό και όχι μακροπροληπτικό. Δηλαδή πρέπει να εξετάζει το σύστημα συνολικά ώστε να αποφύγουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, να βρεθούν σε δύσκολη θέση όλα μαζί ταυτόχρονα. Θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε τη σφαίροντα των ε, καταναλωτών και των φορολογούμενων. Κοιτάξτε τι είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Είδαμε επιτόκια κοντά στο μηδέν. Βρισκόμαστε σε, σε άγνωστους τόπους και μέχρι στιγμή η νομοθεσία που υιοθετήθηκε, υιοθετήθηκε τη στιγμή που προσπαθούσαμε να σβήσουμε τη φωτιά. Ενώ η νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές ώστε να είναι πιο στεναρή. Μάλλον δεν έχουμε κάνει αρκετά για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Και ναι, πράγματι υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες στην τομεακή νομοθεσία. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών διαφορές όσον αφορά την διαφάνεια και τις κυρώσεις. Και συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο οριζόντιο συντονισμό σε αυτές τις πτυχές της νομοθεσίας. Η πέμπτη σκέψη που θέλω να σας παρουσιάσω είναι η ιδέα ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή και τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης. Η ιδέα αυτή είναι επικίνδυνη. Γιατί, διότι υπονοεί ότι υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στην καλή νομοθετική ρύθμιση από τη μία και την ανάπτυξη και, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από την άλλη. Η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως ε, είπε ο Ανδρέα Ένρια, επικεφαλής ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η βασική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ανάπτυξη είναι να μην προκαλέσει ε, οικονομική κρίση. Κοιτάξτε και αυξανόμενο αριθμό μελετών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΣΑ, ε, της BIS κλπ. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι ε, ο υπερβαλλικά μεγάλος χρηματοπιστωτικός τομέας εμποδίζει την ανάπτυξη. Κλείνοντας, να πω ότι τη στιγμή που η πολιτική μεταφέρεται από την ιδέα ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε την μη τραπεζική πιστοτική δραστηριότητα στην ιδέα ότι πρέπει να την προωθήσουμε μέσω της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, είναι όλο και πιο επίγον να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε και πώς θα το κάνουμε αυτό ρυθμίζοντα ε, τη μη τραπεζική πιστοτική δραστηριότητα, τον λεγόμενο σκιώδη τραπεζικό τομέα. Γιατί? Για να διασφαλίσουμε τη ε, ε, δημοσιονομική σταθερότητα και να μειώσουμε το, τον κίνδυνο για τους φορολογούμενους και τους καταναλωτές. Αυτές είναι οι πραγματικές προϋποθέσεις για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι ο πυλώνας της ζήτησης που αποτελεί και ε, την βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, διότι η κατανάλωση ε, αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much ε, to... Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τις τόσο έστοχες παρατηρήσεις σας και για τη συνεισφορά σας στη συζήτησή μας, την αξιολόγηση που κάνουμε και βέβαια ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κάποια αντίθεση, αντίφαση ανάμεσα στην οικονομική σταθερότητα, ρύθμιση και ανάπτυξη. Αντίθετα, εμείς θέλουμε να εντοπίσουμε καλύτερους τρόπους ώστε αφενός να αντιμετωπίσουμε τα κενά στη ρύθμιση και όντως το σκιώδες τραπεζικό σύστημα είναι μια τέτοια περίπτωση, αφετέρου δε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο και τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί ως τώρα και άρα να συμπεράνουμε κατά πόσο βοηθάει στο να έχουμε μια σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Η ισορροπία είναι λεπτή και γι' αυτό είμαστε εδώ ακριβώς, για να μελετήσουμε το θέμα να το εξετάσουμε και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Εδώ δεν πρέπει να διστάσουμε κάθε άλλο. Συγχρόνως, κανείς δεν γνωρίζει συνδυασμένες όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις τι συνέπειες έχουν. Και όσοι νομοθέτες θέλουμε και εμείς να εντοπίσουμε προβλήματα και να βρούμε καλύτερες λύσεις ή δυνατόν. Τώρα, Περνάμε στη συζήτηση στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Και ο πρώτος είναι ο κύριος Βάλς, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βλέπω κατά πρόσωπο γιατί το μικρόφωνο με υποχρεώνει να στρίβω προς την άλλη πλευρά. Ή δεν θα με ακούει κανείς από το μικρόφωνο ή δεν θα μπορώ να σας βλέπω να μην το θεωρήσετε αυτό ότι είναι αγένεια βέβαια από τη δική μου πλευρά. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται στην διάταξη των εδράνων. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχετε έρθει σε αυτή την ακρόαση σήμερα. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό έχει προσπαθήσει να έχει μια συνολική εικόνα για το συνολικό αποτέλεσμα των ε, νομοθετικών μέτρων που έχουν εγκριθεί. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο όπως ξέρετε κι εσείς. Η Κομισιόν έχει αντιμετωπίσει και πολλές δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θεωρούμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις δυσκολίες. Όταν η Κομισιόν θέλει να φτάσει στο σημείο να αποσύρει και νομοθετήματα από το παρελθόν. Είναι απαραίτητο όμως να κάνουμε μια επισκόπηση. Ξέρουμε ότι πολλά νομοθετήματα και άλλες ρυθμιστικές πράξεις επίκυνται επίσης. Αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος μας προηγουμένως. Έχω απλώς περιοριστεί σε ορισμένα θέματα που θα ήθελα να απευθύνω σε όλους σας ή σε συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένα μέλη του πάνελ που με ενδιαφέρουν. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά όλα τα μέλη του πάνελ. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Άμα μιλάμε για ένα απολογισμό, πώς μπορεί αυτός ο απολογισμός, το stock taking, να βελτιωθεί κατά την άποψή σας στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη δική σας άποψη, πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση αυτού του θέματος από την Κομισιόν με μια συνολική μελέτη, γιατί και αυτό θα ήταν κάτι το πολύ σημαντικό που θα μπορούσε να διευκρινίσει καλύτερα τα πράγματα και να μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων όλων αυτών των νομοθετημάτων μέσω μιας μελέτης. Έχω τώρα ένα ερώτημα στον καθηγητή κύριο Μολώνη και τον Γενικό Γραμματέα Άινταν της Finance Watch. Έχετε μιλήσει για τα θέματα των ε, ε, τραπεζικών φορέων και των ασφαλιστικών τομέων, η ΜΕΝ και η ΔΕ. Πού βλέπετε εσείς να υπάρχει δυνατότητα μια συνολικής βελτίωσης στην ε, ρύθμιση ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο τομέα και κατά την άποψή σας πώς ε, αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι δεν συναρμόζονται καλά οι ρυθμίσεις μεταξύ των δύο τομέων, του ασφαλιστικού και του τραπεζικού. Την κυρία Κόλλη και τον κύριο Γκρέλ τώρα. Θα ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε την προστασία του καταναλωτή από τους κινδύνους, ότι δηλαδή εάν θεωρείτε ότι η νομοθεσία αντιμετωπίζει αυτό το στόχο και δεν είναι απλώς μια οικονομική ρύθμιση. Κατά πόσο πιστεύετε ότι υπάρχουν και αρνητικά αποτελέσματα από τις ρυθμίσεις που αφορούν τον κίνδυνο για τον καταναλωτή σε σχέση με τη δραστηριότητα Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πακέτο επενδυτικών μέτρων που θα έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό το ερώτημά μου είναι το εξή. Στον τομέα, στην κυρία Κόλλη και στον κύριο Γκριλ, στον τομέα αυτό μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και πώς θα βλέπατε το θέμα αυτό για τους μικρομεσαίους παίκτες στην αγορά στον τομέα των ασφαλιστικών και στον τομέα των τραπεζικών. Το τελευταίο ερώτημά μου αφορά την πράσινη βίβλο της Κομισιόν για την Ένωση Κεφαλουχικών Αγορών. Η Οικονομική και Νοσηματική Επιτροπή έχει εγκρίνει σήμερα μια ένα ψήφισμα και μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα της ε, ενίας αγοράς κεφαλαίου. Και εδώ μας ε, ενδιαφέρει το θέμα της λειτουργίας της τιτλοποίησης και των φυλαδίων που έχουν να κάνουν με την ε, πρόσβαση σε πληροφορίες των παιδιτών. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες βελτιώσεις ώστε να δώσει μεγαλύτερη όθηση σε αυτή την αγορά και επίσης πώς μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων του χρηματοπιστωτικού τοπίου. Έχω και περαιτέρω ερώτημα, ερωτήματα βέβαια, αλλά δεν θέλω να σας επιβαρύνω με όλα αυτά τα ερωτήματα ομού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βάλς. Ο Πολ Τάγκ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναγνωρίζω κάποια στοιχεία από τις διαμαρτυρίες, από τα παράπονα όσον αφορά την υπερβολική ρύθμιση μετά την κρίση, αλλά και πριν είχα συναντηθεί με τον κλάδο και είχα ακούσει διάφορα παράπονα για τη ρύθμιση και είναι σαφή και από τον, μάλλον και από τον εισηγητή και από τον πρόεδρο. Το θέμα δεν είναι να πάμε πίσω, δεν θα ήταν καλό αυτό. Θέλω. Λοιπόν, στον πρόσωπο των ασφαλίσεων να μας πει κάτι που να μπορεί και εμάς να μας βοηθήσει. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις τράπεζες. Έτσι καλώς ε, δεν είμαστε πολύ δημοφιλείς με τη ρύθμισή μας, αλλά ελάτε να μας πείτε κάτι γιατί αυτό που θέλουμε να ακούσουμε από τον οικονομικό τομέα είναι ότι δουλεύουμε προς το συμφέρον του κόσμου. Και τότε να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε στο χρηματοποστοτικό τομέα. Το θέμα δεν είναι να λέμε συνέχεια απασχόληση. Δεν πρόκειται για να κάνουμε πίσω σαν αφορά τη ρύθμιση. Θέλουμε όμως από εσά να ακούσουμε τι θέλετε να κάνουμε ώστε να φανεί ότι εσείς εξυπηρετείτε τον κόσμο και ότι δουλεύετε κι εσείς και οι τράπεζες προς το συμφέρον του κόσμου. Έχω μια ερώτηση. Ερωτήσεις θέλω να κάνω γιατί νομίζω ότι είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να κάνουμε τις ερωτήσεις και μετά να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τον κύριο Νάιντεμ, Δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς. Έχω μια ερώτηση προς αυτόν και προς τον κύριο Μαλώνη. Διότι μίλησαν για προστασία του καταναλωτή, χωρίς να διευκρινίσουν. Θα ήθελα να το καταλάβω περισσότερο, γιατί αυτό με έκανε μένα να σκεφτώ ότι εσείς βλέπετε τρόπους για να βελτιωθεί η προστασία του καταναλωτή. Μπορεί να είναι στη φαντασία μου βέβαια, αλλά θα ήθελα να το ξέρω. Σαν να λέτε ότι δεν ασχοληθήκαμε αρκετά με τον καταναλωτή στην κρίση αυτή. Τι δυνατότητες βλέπετε εσείς. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Μπορούμε να έχουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων ίσως. Σύντομα, αν μπορείτε. Δύο, Τρία λεπτά ο καθένας σας. Ποιος θα αρχίσει? Παρακαλώ. Ο κύριος Νάιτσον. Νίσνταμ προφέρεται. Είμαι Γάλλος, παρότι το όνομά μου είναι ε, Ολλανδικό. Θα συμφωνήσω βεβαίως με τον κύριο Μπάλτσο ότι φυσικά μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο, μάλιστα οφείλουμε να δούμε τον αντίκτυπο ε, των ε, ρυθμίσεων και των νομοθετημάτων, αλλά το κακό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες πλέον. Ας πούμε, ε, στο RD4 βλέπετε ότι δεν θα υλοποιηθεί πριν από το 2019 ε, και μάλιστα δεν έχουν ε, οριστεί ακόμα ούτε καν όλες οι λεπτομέρειες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ποσοστοποιήσουμε το κόστος ε, μιας ε, κρίσης. Εάν δει κανείς ε, την μελέτη αντικτύπων πόσο θα κοστίσει αυτό ας πούμε σαν κόστος συμμόρφωσης στην τράπεζα, αυτό είναι το εύκολο και εγώ μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε τόσο κόσμο και θα κοστίσει τόσο. Αλλά το κόστος για την κοινωνία μιας τέτοιας κρίσης είναι σαφώς μεγαλύτερο και αν θέλετε να κάνετε μια πραγματική μελέτη αντικτύπων που θα πρέπει να δείτε όλες τις πλευρές. Επίσης να μην λησμονούμε ότι αυτή η κρίση είναι το αποτέλεσμα της απορρίθμισης, deregulation και όχι της ρύθμισης, regulation. Να μην ε, προχωράμε λοιπόν σε λάθος διάγνωση. Ε, στην αξιολόγηση βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε και το πρόβλημα ενός μιας τάσης πληρωμών, default, ή το πόσο μακριά είναι το ενδεχόμενο ενός default. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Ε, Κέλλερ. Θα ήθελα εδώ να παραθέσω τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς, ο οποίος είπε ότι ίσως θα πρέπει ε, ε, να δούμε πότε θα πρέπει να κάνουμε τις μελέτες ατικτύπου τις οποίες κάνουμε συνήθως στην αρχή, αλλά όχι στο τέλος. Ίσως, ίσως λέω, θα πρέπει να κάνουμε στο τέλος μια μελέτη για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος στο τέλος της ολοκλήρωσης διαδικασίας. Ε, ο κύριος ε, ε, νίσταμε είπε κάτι πολύ σωστά σε σχέση με το κόστος και το όφελος του, των κανονιστικών ρυθμίσεων. Στην Insolvency 2 δεν έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, αξιολογήσεις ή εκτιμήσεις ε, κόστου. Πάντως και ο κλάδος και οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι για την εφαρμογή του Solvency 2 θα έχουμε ένα κόστος περίπου 4,2 δις ενώ το κέρδος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Όσον αφορά τώρα το τι κάνουμε όταν βλέπουμε ε, τους ε, κινδύνους και ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία να πω ότι μας ζητούν να δούμε ας πούμε ορισμένα στοιχεία της Solvency 2 ε, και δεν κάνουμε μια έτσι, λεπτομερή βαθμονόμηση ε, χωρίς να λαμβάνουμε καθόλου υπόψη βέβαια τους κινδύνους. Απλώς εμείς ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που είναι εγγενείς στην οικονομία. Βεβαίως προκύπτει ένα ζήτημα ότι ναι, δεν έχουμε ακόμα ένα μοντέλο στις ασφάλειες ζωής που να είναι πραγματικά πλήρες. Επίσης και ένα άλλο ζήτημα μέσω του, της πράσινης βίβλου, μια και την αναφέρατε, είναι να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή τάξη ε, για τις ε, επενδύσεις ε, και ένα τελευταίο, νομίζω ο κύριος Τάγκ ρώτησε, μπορείτε να, είπε, μπορείτε να μου κάνετε μια συγκεκριμένη πρόταση ε, που, ε, που να δείχνει ότι θα βοηθήσουν οι αλλαγές ε, του κανονισμού. Ε, κοιτάξτε, όταν δει κανεί τη δέσμη των ε, κανονισμών που μας έχουν έρθει, ε, και που μελετούμε πρέπει να πούμε ότι καταλήγουμε στο ότι έχουμε λιγότερες, ε, λιγότερους κινδύνους ε, για τους με μεμονωμένους ανθρώπους. Ε, εμείς ε, δεν έχουμε ένα ειδικό ε, μοντέλο για τις απλές περιπτώσεις. Θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο το οποίο να λαμβάνει υπόψη και τα assets και τις liabilities και τα θετικά και τα αρνητικά και τις υποχρεώσεις. Επομένως, στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κλάδος δίνει ε, αυτή τη στιγμή κίνητρα για οτιδήποτε δεν είναι απολύτως ή δεν φαίνεται απολύτως εγγυημένο ε, και, ε, και όλο και περισσότερο πηγαίνουμε προς νέα, νέες επενδύσεις που είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένα προϊόντα. Και εκεί είναι το ζήτημα να βρούμε ποια είναι τα πιο ασφαλή και τα πιο κατάλληλα προϊόντα για να συνδεθούν με τις ε, συντάξεις ε, και πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν ε, θεωρούμαστε traders ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα ψηλές διακυμάνσεις και επομένως για μας το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το default. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σύντομα για την προστασία του καταναλωτών, διότι δεν είχα καταλάβει ότι πρέπει να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα. Να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας τρεις παρατηρήσεις. Η στοχευμένη βελτίωση στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα των καταναλωτών να συγκρίνουν μεταξύ τους τα προϊόντα και να καταλάβουν πού επενδύουν. Άλλες δύο παρατηρήσεις. Ε, στο CMU. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ε, επενδυτών λιανικής, των μικρών επενδυτών και τέλος, εάν μεταφέρουμε μέρος του κινδύνου από τις τράπεζες στα, στα εξωτερικά ταμεία μπορούμε να αυξήσουμε τον ηθικό κίνδυνο. Σας ευχαριστώ και το συγγνώμη που δευτερολόγησα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις ερωτήσεις σας. Ε, να είμαι σύντομη όσον αφορά την μελέτη επιπτώσεων. Νομίζω ότι είναι πράγματι κρίσιμη να κάνω τέσσερις μικρές προτάσεις. Καταρχάς, να γίνει μια πιο δυνατή προσπάθεια να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά ε, θα υπάρχουν έτσι διάφορες προοπτικές ε, στην όλη διαδικασία. Και δεύτερον, benchmarking, να έχουμε σαφή σημεία αναφοράς ώστε να μπορέσουμε σε τρία ή πέντε χρόνια να ξανααξιολογήσουμε την επίτευξη των στόχων. Ε, και τέλος, ε, οι προθεσμίες, τα προγράμματα δηλαδή, ε, να μοιραστούν σε διάφορες περιόδους τριών-πέντε ετών. Και τέλος, να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να προβλέψουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν το πώς η νομοθεσία επηρεάζει τις αγορές. Επίσης, όσον αφορά τα διατομεακά θέματα και την ερώτηση που τέθηκε, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει δουλειά πάνω στις κυρώσεις, επίσης στις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών που διαφέρουν και επίσης όσον αφορά την ισοδυναμία και την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Ε, υπάρχουν Στην ευρωπαϊκή αγορά υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Παραδείγματα όπου τα πράγματα ίσως να μην ταιριάζουν με το σύστημα του παρελθόντο. Ε, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων. Έχουμε πληροφορίες που έρχονται από διάφορες ε, πηγές ε, και η αίσθηση μου είναι ότι το πρόγραμμα άρχισε να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο με όλο και περισσότερες διαφορετικές αποχρώσεις. Παρότι δεν θέλουμε να ανακαλέσουμε τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να μάθουμε ένας από τον άλλον. Το ε, AIFND ε, βλέπει με συγκεκριμένο ρόλο το θέμα της ε, διακυβέρνησης. Είχαμε διάφορες προτάσεις. Μπορεί απομονωμένε οι προτάσεις αυτές να λειτουργούν πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς συνδυάζονται μεταξύ τους και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα συστήματα. Και τέλος, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει εδώ ανάγκη να υπάρχει συνέπεια. Στο MIFID 2, για παράδειγμα, βλέπουμε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τις ε, παρεμβάσεις ε, για τα προϊόντα και, την, και το σχεδιασμό των προϊόντων. Είναι απαραίτητοι αυτοί, αυτοί οι κανόνες. Από την άλλη μεριά όμως, στην Ένωση Κεφαλαιογρών βλέπουμε ότι αυξάνουμε ε, το κατόφλι για τα προσπέκτους, το οποίο σημαίνει ότι ίσως να διευκολύνουμε την πρόσβαση επικίνδυνων εκδοτών στην αγορά. και θα πρέπει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία να εξετάσουμε ποιος είναι ο καταναλωτής. Ας εξετάσουμε πάλι τους ορισμούς μας, ας εξετάσουμε πάλι ε, τα κατόφλια, τις κατώτατες τιμές, ε, ποιους θέλουμε να ενθαρρύνουμε και ποιους θέλουμε να προστατεύσουμε. Για να αποφύγουμε αυτές ε, τις πιθανότατα μεγάλες ασυνέπειες στο συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις μελέτες επιπτώσεων, Πολλά ήδη υπόθηκαν, θα ήθελα όμως να προσθέσω το εξής. Θα πρέπει να έχουμε μία συνολική αξιολόγηση. Θα πρέπει να έχουμε μία συνολική επισκόπηση. Τι κάνει το Κοινοβούλιο, το, η Κομισιόν, τι μέτρα έχουν λάβει οι νομοθέτες σε τοπικό επίπεδο Και επίση αυτό που ανέφερα πριν, το οποίο μπορεί να αποτελεί σημαντικό κινδύνο για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 20 με 30% του συνολικού κεφαλαίου ε, όπως μου είπαν χθε ε, με email ε, μπορεί να ε, διαγραφεί όσον αφορά τα κεφάλαια των τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο κίνδυνος ε, θα είναι τελικά οι τράπεζες να πρέπει να αποσυρθούν από κάποιους τομείς ε, και ένας ιδιαίτερα ευάλωτος τομέας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι πιθανότατα να μην είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να λάβει κανείς αποφάσεις σχετικά με την χορήγηση δανείων και έτσι οι τράπεζες μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν το δανεισμό στον τομέα αυτών ή να ε, ε, εξαναγκαστούν ε, να συγχωνευτούν και δεν ξέρω εάν μας συμφέρει να έχουμε πιο πολλές μεγάλες τράπεζες και λιγότερες μικρές και περιφερειακές τράπεζες. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Η Κέιτ Σουίνμπορν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε διαφορετικέ απόψει και διαφορετικού οικονομικού τομεί που καλύπτονται εδώ. Είναι πολύ δύσκολο με δύο μονάχα σύντομε ερωτήσει να φτάσει κανεί στην ρίζα μερικών από τα βασικά ερωτήματα που έχουμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτή τη επισκόπηση. Θα ήθελα όμω πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσω αυτό το οποίο ε, είναι στην ατζέντα του κύριου Τίμερμανς. Είπε ότι ο κάθε τριγωνικός διάλογος έχει τις δικές του συμβαστικές λύσεις υπάρχει τόσο μεγάλη εστίαση στο να υπάρχει μια συμβαστική λύση που τελικά δεν έχει κανείς μια συνολική εικόνα για το πώς αυτή η συμβαστική λύση συνδέεται με τις άλλες. Θα ήθελα λοιπόν να έχω μια, ε, την άποψή σας για θέματα όπως το IMD2 για τις ε, ασφαλιστικές υπηρεσίες που έχει πολλά ερωτήματα ακόμα που είναι ανοιχτά και επίσης για τα πρόσθετα το πρόσθετο άκτος που δημιουργείται με τα κεντρικά αποθετήρια για τα παράγωγα. Πώς λοιπόν μπορείτε να βρείτε συνδέσεις μεταξύ των ε, διαφορών τομέων. Φυσικά υπάρχει η ανάγκη παράδοσης αναφορών που έχει αυξηθεί σημαντικά. Σωστό είναι αυτό. Καλό είναι να έχουμε πληροφόρηση προς τους πελάτες. Αυτό έχει γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο με τις δεσμεύσεις των G20. Αλλά είδα ένα διάγραμμα τύπου VEN από ένα, μια εταιρεία συμβούλων και παρουσιάζαν το CSTR και το MIFID που δεν ήταν συνδεόμενα διαγράμματα, ήταν διάφορες νησίδες που είχαν μια πολύ ε, αμυδρή διασύνδεση μεταξύ τους. Πώς θα αριθμίσετε αυτό το πρόβλημα και πώς θα εξασφαλίσετε ότι είναι πιο τυποποιημένη η μεθοδολογία σε αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και επίση υπάρχουν και οι μη νομοθετικέ λύσει που ανέφερε η κυρία Μαλόνι υπό τη μορφή τη αλλαγή νοοτροπία. Είδαμε την επισκόπηση του ΕΒ για τι δίκαιε και αποτελεσματικέ εταιρείε που βασίζεται κυρίω στην προσωπική ευθύνη του καθένα ο οποίος συμμετέχει στην παραγωγή αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Πόσα από αυτά λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μονάχα σε ένα εθνικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης για τα χρηματοοικονομικά συμβούλια. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα του καταναλωτή και συγκεκριμένα του συνταξιούχου, κάποιος θα πρέπει να λάβει την ευθύνη για το μέλλον τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονάχα ευρωπαϊκό κράτος το οποίο θα μπορεί να δώσει στους συνταξιούχους μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πώς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό περιβάλλον για να συμβάλλουν και οι συνταξιούχοι στους τομείς αυτούς ώστε να έχουν ε, μακροχρόνια ένα σημαντικό κομπόδεμα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μετά τη σύνταξη. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος ταιριάζει καλά, δεν είναι πια εδώ. Ο Μίγκελ Βιέγκς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα να υπάρχουν κάποια παράπονα σε σχέση με τα υπερβολικά τέλη που υπερβάλλονται στους, ε, σε του τομέα και κάποιες ε, διαμαρτυρίες σε σχέση με την υπερβολική ρύθμιση και τις υπερβολικές απαιτήσει από το ρυθμιστικό τομέα. Είναι καλό να θυμηθούμε ότι το κόστος και το, βάρος που έφερε η κρίση στους ώμους των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν καν αξιολογηθεί πλήρω, αλλά κυμαίνονται γύρω στο 40% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επομένως, αν υπάρχει μια θεμητή, θεμητό παράπονο σε σχέση με τα αποτελέσματα της κρίσης, νομίζω ότι οι καταναλωτές πρέπει να διαμαρτύρονται και όχι οι τραπεζίτες. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι το εξή ενώπιον της κρίσης, ενώπιον της ανάγκης να ξεπεράσουμε την ανικανότητα των αγορών να αυτορυθμιστεί, να αυτορυθμιστούν και να λύσουν τα προβλήματα. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προχωρήσουμε προς μια ρύθμιση η οποία μπορεί να είναι πολύπλοκη αλλά είναι και απαραίτητη. Αν υπάρχει λοιπόν η γενική συμφωνία ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, αναρωτιέμαι και σας θέτω το ερώτημα αν μπορεί να είναι θεμητή αυτή η διαμαρτυρία για την ε, υπερβολική ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη τα ολέθρια αποτελέσματα που είχε η κρίση στην κοινωνία μας και την οικονομία μας. Για την διαδικασία αυτή καθεαυτή πιστεύω ότι θέτει μια σειρά ερωτημάτων για τα οποία θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την άποψη των καλεσμένων μας. Για το Ταμείο Επίλυσης και Ανάκαμψης κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι είναι ελάχιστο το ποσό του ταμείου αυτού σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθεί ο τραπεζικός τομέας. Είναι στα γόνα το ωκεανό τα 55 αυτά δισεκατομμύρια και η απάντηση που μας δίνεται είναι ότι είναι λίγα τα λεφτά αυτά γιατί μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ γιατί η εποπτεία θα είναι επαρκής και υπάρχουν οι τράπεζες οι οποίες είναι όπως λέμε, too big to fail, πολύ μεγάλες για να αποτύχουν, οι οποίες δεν κινδυνεύουν. Επίσης υπάρχει, ε, υπάρχουν ορισμένα θέματα που αφήνει κατά μέρο η τραπεζική εποπτεία. Υπάρχει το θέμα του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των τραπεζών. Υπήρξε μια έκθεση η οποία ζητούσε την, ε, το διαχωρισμό μεταξύ των επενδυτικών δραστηριοτήτων και των φυσιολογικών, των συνηθισμένων ε, τραπεζικών δραστηριοτήτων. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν αυτό το ερώτημα σας φαίνεται ουσιαστικό, μήπως είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ της κανονικής τραπεζικής και της επενδυτικής και δοσκοπικής δραστηριότητας με στόχο να προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές και τους καταθέτες και να εμποδίσουμε ότι οι τράπεζες τσογάρουν τα χρήματα τα οποία καταθέτουν οι καταναλωτές. Το άλλο θέμα είναι το σύστημα των σκιωδών τραπεζών, το shadow banking, που είναι αυτή τη στιγμή το ίμιση του ενεργητικού του συνολικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει ξεπεράσει το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την κρίση. Ποια είναι η άποψή σας και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τις, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι η αιτία της κρίσης ή αποτέλεσμα της κρίσης. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί για το αν θα πρέπει και στην περίπτωση του σκιωδό συστήματος θα πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος για τους ισολογισμούς και την διαφυγή από τη ρύθμιση. Επίσης υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της ανάγκης να υπάρξει στάθμιση κινδύνου για τα κεφάλαια και της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο οι κεφαλουχικές απαιτήσει είναι αυτό ακριβώς που εμποδίζει τις τράπεζες να μην δανείσουν τους τομείς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προτιμούν να αγοράσουν απλώς κρατικά ομόλογα. Το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με τη φορολογία. Όπως γνωρίζετε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικά πληρώνει περιορισμένους φόρους. Έχει πολύ χαμηλό επίπεδο φορολογίας, πολύ πιο χαμηλό από οποιαδήποτε από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε όλες τις ε, δραστηριότητες φόρο και φοροδιαφυγής που σήμερα είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η άποψη των καλεσμένων μας για το κατά πόσο ο τομέας αυτός πράγματι συμβάλλει σήμερα στο να αντιμετωπιστεί αυτό το ηθικό θέμα και να εξασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα πληρώνει το τμήμα των φόρων που του αντιστοιχεί όπως σε οποιοδήποτε πολίτη και επίσης για το κατά πόσο πράγματι συμμετέχουν σε όλα τα μέτρα διαφάνειας για να αποφευθεί η μεταφορά κερδών σε φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ απαντήσεις σε αυτό το γύρο ερωτήσεων. Ποιος θα αρχίσει τώρα, ο κύριος Γκρόου, Finance Watch. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την ερώτηση της κυρίας Σουίνμπερτ όσον αφορά τις προδιαγραφές πληροφοριών αναφοράς μεταξύ τεσσάρων ε, νομοθετικών οργάνων είναι ε, μια, ένα εγχείρημα που όπως είπα και στην αρχή αρκετά δύσκολο. Για το κατάλληλο περιβάλλον όσον αφορά τους καταναλωτές και το μέλλον, οι βιώσιμες επενδύσεις είναι το βασικό γιατί αποφέρουν χρήματα. Όχι απαραίτητα αυτό που προβλέπετε τώρα στο σχέδιο CMU που προβλέπει εύκολο κέρδος για να αποφύγουμε την κατάρρευση, την πλήρη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι τράπεζες χρειαζόντουσαν ρευστότητα. Κανένας δεν ήθελε βέβαια να καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέπειο όμως αυτού είναι να έχουμε μηδενική ανάπτυξη. Οπότε ουσιαστικά βρισκόμαστε στην χειρότερη περίοδο οικονομικά που γνωρίζουμε τους τελευταίους δύο αιώνες. Η κύρια ανησυχία του κόσμου δηλαδή είναι μηδέν επιτόκια για να αποφύγουμε την κατάρρευση του συστήματος. Αν οι επόμενοι σταξιδοτούμενοι θέλουν περισσότερα κέρδη, πρέπει να αναλάβουν και μεγαλύτερους κινδύνους. Το θέμα όμως είναι ότι ως κοινωνία δεν πρέπει να περάσουμε τον κίνδυνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τους καταναλωτές αν οι καταναλωτές δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να συγκρίνουν κινδύνους και να παίρνουν αποφάσεις. Συνεπώς, πρέπει να εισάγουμε κάποιου είδους παράγοντα ηθικού κινδύνου. Το στεξιδιωτικό ταμείο που κινδύνεψε περισσότερο ήταν ιδιωτικό. Αυτό λοιπόν είχα να πω για να απαντήσω στην κυρία Σίνμπερτ. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση του κ. ναι, συμφωνώ ότι τα 55 δις, το ταμείο δηλαδή εξυγένσης με αυτό το κεφάλαιο, όντως δεν φτάνει, οι too big to fail δεν καλύπτονται, το ξέρουμε, το έχουμε σκεφτεί. Το bail-in λειτουργεί έτσι καλλιώς μόνο για μικρές τράπεζες, όπως έγινε στην Κύπρο το Μάρτιο του 2013. Δεν θα λειτουργήσει για μεγάλες τράπεζες σε ένα Σαββατοκύριακο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα σχέδια διάσωσης των μεγάλων ε, τραπεζών είναι 1800 σελίδες. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρόλ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σύντομα και εγώ σε αυτό που ρωτήσατε όσον αφορά τις απαιτήσει αναφοράς και πληροφοριών. Όντως πρέπει να είναι κάτι λογικό και να υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στις μεγάλες τράπεζες και τις πιο μικρές με λιγότερο περίπλοκα συστήματα. Δεν ξέρω τι πηγές χρειάζονται αρμόδιες αρχές για 15 εκατομμύρια με καθημερινές συναλλαγές δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα καν να απορροφήσουν τόσες πολλές πληροφορίες. Πάντως για τις πιο μικρές τράπεζες το reporting αυτό πρέπει να είναι σε τέτοιο μέγεθος που να μπορούν να το αφομοιώσουν εύκολα. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή τις ίδιες προδιαγραφές ενημέρωσης στις μικρές και στις μεγάλες τράπεζες. το Ταμείο Επίλυσης, Διάσωσης, ναι φυσικά δεν θέλουμε να πληρώνουμε δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Δεν θέλουμε δηλαδή να συνεισφέρουμε στο Ταμείο αυτό διάσωσης και στα εθνικά, στο κρατικό δηλαδή προπολογισμό συγχρόνως, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι φορολογούμε δύο φορές. Η φόρη εξάλλου των τραπεζών σε μια κανονική χρονιά και μιλάω από τη δικιά μου βέβαια την πλευρά, είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι πληρώνουν οι ιδιώτες. Τέλος, για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, ναι, πρέπει να ρυθμιστεί, σαφώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι άδικο αν έχουν τις ίδιες δραστηριότητες, χωρίς όμως ρύθμιση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Κέλλερ. Ναι, όσον αφορά την ερώτηση της ε, κυρίας Σούμπερν, ε, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα ε, σχετικά με τη δημοσίευση του κόστους και των χρεώσεων. Έχουμε το άρθρο 3 το οποίο λέει ότι θα πρέπει να ε, δίνονται από, από, από την ασφαλιστική εταιρεία ε, ε, συγκεκριμένα στοιχεία και επίσης έχουμε και το άρθρο 22.3 όπου αναφέρονται ότι τα κόστη και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με συνολικό τρόπο δηλαδή περίπου το ίδιο πράγμα λέει αλλά με διαφορετική διατύπωση ε, δηλαδή θα πρέπει ο, ο, ο, ο υπεύθυνο να ε, σκεφτεί με ποιο τρόπο θα ε, μπορούσε να παρουσιάσει αυτού του είδους το κόστος, αλλά στην ουσία μπορεί να κάνει, για μια απλή λύση, μπορεί να κάνει μια παραπομπή στο δεύτερο κανονισμό που ανέφερα. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, πρέπει να σας πω ότι τώρα φύγαμε από τη Solvency 1 και πηγαίνουμε πλέον στη Solvency 2 Έχουμε 71 reporting templates πλέον, αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά υπάρχουν και επιπλέον ε, υποχρεώσεις που μας έχουν επιβληθεί στον τομέα της, των ασφαλιών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εν τέλει μετά από μακρές συζητήσεις ανάμεσα στην ΑΙΟΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, νομίζω ότι τώρα πλέον έχουμε ένα σωστό πλαίσιο ε, και ε, στην ουσία δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις απόψεις της ΑΙΟΠΑ. Αλλά έγινε πολλή συζήτηση και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά σχόλια. Όσον αφορά ε, τις ε, υποχρεώσεις ε, αναφορών reporting requirements. Βεβαίως είναι, δεν είναι κάτι σταθερό που δεν μπορεί να αλλάξει. Αντιθέτως πρόκειται για μια διαδικασία bottom-up και πιστεύουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συζητούν έτσι ώστε να βρουν τον τρόπο της αναφοράς που περισσότερο τους ταιριάζει. Οι παρόντες ε, κανονισμοί μπορούν να έχουν και στα πλαίσια του ESM ε, ε και ε, γενικότερα μπορούν να έχουν μερικά θετικά στοιχεία. Πιστεύουμε ότι ίσως ε, ο κανονισμός δεν δεν, δεν αφορά ούτε καν το 50% του μηχανισμού που θα χρειαζόταν για πραγματική εποπτεία της ε, αγοράς. Ε, νομίζω ότι είναι η, η, η λυπηρή πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα όπως η liability ή όπως οι εγκληματικές πράξεις, ε, ε, οι υποχειρήσεις της αγοράς ε, κλπ που είναι πολύ σημαντικά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ε, μπορεί κανείς να δει πώς ε, εφαρμόζουν τους, τις κυρώσεις ε, τα διάφορα κράτη-μέλη, πώς μπορεί να συγκρίνει κανείς τις κυρώσεις. Και τέλος ένα τελικό σχόλιο για την Τραπεζική Ένωση. Ναι, επειδή υπάρχει κίνδυνος αρμπιτράζ, είναι γεγονός ότι είναι σημαντικό να δει κανείς ε, την κατάσταση στα πλαίσια όμως ε, και της, της παγκόσμιας ε, κατάστασης καθώς επίσης και σε σχέση με τα αυτά που προβλέπει και το Stability Board. Ο Μάρκος Δάνη, έχουμε δυνατότητα να πάρουμε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Παρακαλώ. Όσοι συνάδελφοι θέλουν ε, να σηκώσουν το χέρι τους να πάρουν το λόγο, Σβάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Συμφωνώ με αυτό που υπονόησαν αρκετοί ομιλητέ ότι η χρηματοπιστωτική νομοθεσία δεν είναι πιο αποτελεσματική αν είναι περισσότερη. Δεν εξαρτάται δηλαδή από τον όγκο. Ο αριθμό σελίδων, ο αριθμό ε, οδηγιών, κανονισμών, ε, κατευθυνότηση πράξεων, ο όγκο που παράγουμε δεν είναι μέτρο για να ε, υπολογίσουμε αν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μα ή όχι. Άκουσα βέβαια κάποιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομιλητών. Μερικοί θέλουν συγγύρισμα, μερικοί όχι τόσο πολύ. Όσοι είναι υπέρ πιο ισχυρού νομοθετικού πλαισίου φοβούνται ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρήσουμε τα πρότυπα, εάν συγκυρίσουμε την κατάσταση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα αποτελέσει ευκαιρία για να απαλλαγούμε από κάποια από τα πρότυπα, τα οποία είναι μάλλον ενοχλητικά. Αυτή είναι μια μάλλον τοξική συζήτηση και παραπλανητική. αλλά θα ήταν ενδιαφέρον για μένα να ακούσω κάποια αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με το αν έχουμε πετύχει ή όχι. Τι εννοώ όταν λέω ε, αντικειμενικά κριτήρια. Οι καταναλωτές παίρνουν ε, μεγαλύτερο μερίδιο των χρημάτων, του κέρδους ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Είπατε ότι οι επενδυτές χρειάζονται το εισόδημα αυτό ε, για το μέλλον, για να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους. αλλά μήπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας ε, παίρνει υπερβολικά μεγάλο μερίδιο των χρημάτων που παράγει ο τομέας αυτός. Παράδειγμα, έχουμε το σύστημα της Σουηδίας, όπου οι συντάξεις βασίζονται σε κεφάλαια που δεν βασίζεται όμως ε, στον ακριβό ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. το κόστος ε, για το κεφάλαιο ύψους 0,2% θα μπορούσε να προταθεί για τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια. Δεύτερον, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κανονισμού για την αφαιρεγκαιότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρά τις προσπάθειές μας φαίνεται ότι οι επένδυτες στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές θεωρούν ότι είναι ασφαλής επένδυση. Ότι ιδιαίτερα ο τραπεζικός τομέας είναι ε, ασφαλής επένδυση. Φαίνεται όμως ότι έχουν αυξηθεί τα περιθώρια και ότι θα υπάρχει πρόβλημα ευθύνη ε, στο μέλλον και θα πρέπει ο φορολογούμενος ε, τελικά να πληρώσει. Τι προτείνεται λοιπόν για να λειτουργήσει το πλαίσιο, διότι για μένα αυτό θα αποτελούσε αντικειμενικό κριτήριο. Τέλος, πώς βρίσκεται την ιδέα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βίβλος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από την ε, τομεακή ε, νομοθετική ρύθμιση και να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα ε, επικαλύψεων και αναλογικότητας που δημιουργήσαμε με το καθεστώς που δημιουργήσαμε, όπου έχουμε 40 διαφορετικά νομοθετήματα, ώστε τουλάχιστον όσον αφορά τους ορισμούς, την υποβολή εκθέσεων, για παρόμοιες περιπτώσεις να έχουμε παρόμοια ή κατά προτίμηση όμοια ρύθμιση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις προτάσεις σας και το πώς εσείς ε, αξιολογείτε την, ε, τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Να θέσω εγώ τότε μία ερώτηση προς τον κύριο Γκρουλ. Μήπως θα μπορούσατε να αναπτύξετε αυτό που είπατε για το IFRS. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω συγκεκριμένα σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια, ότι δεν υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στον πυλώνα 1 και 2. Πιστεύετε ότι δεν αξιολογείται σωστά ο κίνδυνος και ότι δεν ενθαρρύνεται η χρηματοδότηση της πραγματική οικονομίας. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να αναπτύξετε περισσότερο το θέμα αυτό. και σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του. Παρακαλώ. Όσον αφορά το IFRS, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Κύριε Πρόεδρε, όσο έχει το σύστημα σήμερα, νομίζω ότι είναι έφεπτο και ότι μπορεί να εφαρμοστεί από τις τράπεζες, όπως είπα και πριν. Υπάρχει μεγάλος φόβος διότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη αντικτύπου σχετικά με το ένα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω η Επιτροπή σας έχει μια υποομάδα που ασχολείται με το θέμα αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ η εφαρμογή στην πράξη που φυσικά είναι επαχθής και απαιτεί, χρόνια, αλλά πέρα από τις κεφαλαιακές απαιτήσει. θα υπάρχει και σημαντικός αντίκτυπος, για, ένας επιπλέον σημαντικός αντίκτυπος για τα κεφάλαια κάτι που θα έχει επιπτώσει και στον δανεισμό και θα δημιουργήσει αστάθεια που πάντα αποτελεί πρόβλημα όταν ε, μιλάμε για ε, την αξιολόγηση της ε, χρηματοοικονομικής κατάστασης. Η σύστασή μας λοιπόν θα ήταν όταν ληφθεί η απόφαση για το ένα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να εξεταστεί συνολικά το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσει, παραμένει ασαφές το πώς ε, κάποια μπάφερ όπως ε, το συστημικό θα εφαρμοστούν στο σύστημα που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από το σώμα των ελεγκτών την προηγούμενη εβδομάδα η Αυστρία ανακοίνωσε ένα τέτοιο μπάφερ και είχε πολύ, είχε πολλές ε, αντιδράσεις. Ε, θα εκτιμούσαμε λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Γκίνγκολτ για το ερώτημά του και επί τη βάση και τη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα συνταξιδετικά ταμεία πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε πιο ρεαλιστές σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να σκεφτείτε για ένα εγχείρημα μακρόπνο, αλλά αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικές εταιρείε έχουν σε πολλές αγορές την δυνατότητα να ανταλλάξει, δηλαδή να ε, γυρίσει πίσω την ασφαλιστική, το ασφαλιστικό συμβόλαιο και να πάρει πίσω τα λεφτά του. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν οι εταιρείε τη δυνατότητα να κάνουν μακροχρόνιε επενδύσει. Βέβαια θα υπάρξουν λύσει μέσα στην Ένωση για τι κεφαλαιοχικέ αγορέ. Θα υπάρξει ίσω μια λύση, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη μία πλευρά. Δεν μπορείτε να ζητάτε να κάνουμε το α, αλλά να διατηρήσουμε συγχρόνω β, μια πλήρη ευελιξία. Θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη λοιπόν αντιμετώπιση για το σημείο αυτό. Και επίση για το, την Ευρωπαϊκή Βίβλο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε που αναφέρατε. Πολλέ φορέ αυτό στρέφεται εναντίον τη δυνατότητα επιλογή προϊόντων. Αν όλοι πάνε προ την ίδια κατεύθυνση, αν όλοι θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τότε χάνεται η δημιουργικότητα που μπορεί να υπάρχει στον τομέα αυτό. Παραδείγματο χάρη, δεν υπάρχει δυνατότητα για μια ασφαλιστική εταιρεία να υπογραμμίσει ποια είναι τα κεφαλογικά αποθέματα που έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να δείξουν ότι αυτό συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ασφαλιστικός τομέας. Πιστεύω γενικά ότι από την οπτική γωνία των ασφαλιστικών εταιριών είναι ότι αν κάποιος ε, αναγκάσει τον κόσμο να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, με νέο τρόπο, αυτό θα οδηγήσει και σε περισσότερους κινδύνους και σε μια κοπαδική αντιμετώπιση και συμπεριφορά, ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ποικιλία στη συμπεριφορά και ο ασφαλιστικός τομέας έχει μείνει στην αγορά <clears throat> όταν πολλοί άλλοι έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Θέλετε να δώσετε λοιπόν στον τομέα αυτό κίνητα για να λειτουργεί διαφορετικά και αυτό σημαίνει πρέπει να έχετε και διαφορετικού κανόνε μερικέ φορέ για να το ενισχύσετε αυτό. Ο καθηγητή Μόραλη. Εγώ συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σα με την ιδέα του να έχουμε αντικειμενικά κρατήρια τα οποία να βασίζονται στην εμπειρία του καταναλωτή και μία από τι σημαντικέ εξελίξει στον τομέα αυτό είναι οι νέοι κανόνε στη μη για την ευκυβερνησία των προϊόντων αν μπορεί να λειτουργήσει αυτό με τους επόπτες να εξετάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανάπτυξη των προϊόντων στον τομέα αυτό και το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο για την παροχή κινήτρων για να έχουν τα οποία είναι θετικά για τους καταναλωτές και δεν είναι απλώς πηγή εισοδήματο. Επανέρχομαι λοιπόν στην ανάγκη εποπτείας και της σωστής εποπτείας για να το εξασφαλίσουμε αυτό για ένα απλό αποταμιευτικό προϊόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αναγνωρίσω. Αλλά είναι ακριβώς το, ίδιο, το είδος ενός σχεδίου που θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτό η Ευρώπη. Έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα σε άλλους τομείς. Αλλά θα πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια φοβάμαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να αναπτύξει απλά προϊόντα και θα ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά θα είναι κάτι πολύ σημαντικό να μπορέσει να επιτευχθεί. Για να υπάρχει μια βίβλος τώρα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για να υπάρχει ένας κοινός κώδικας ε, ορισμών σε σχέση με τις υποπτικές αρχές, τα προϊόντα όπως παράγωγα κτλ. Η δική μου εντύπωση είναι ότι είναι τόσο μεγάλη η πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού πιστωτικού τομέα που αντί να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο <clears throat> θα είναι το επικρατούν σύστημα, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ενιαίες πρακτικές. Αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαμε να έχουμε εναρμονισμένες προσεγγίσεις και κοινού ορισμούς για τα κέρια θέματα που μας απασχολούν. Και εγώ να απαντήσω δεν πιέζω για περισσότερη ρύθμιση, όχι. Πιέζουμε για πιο απλή αλλά πιο ισχυρή ρύθμιση. Είμαστε υπέρ της μόχλευσης για τα επίπεδα solvency. Τώρα για τα τυποποιημένα προϊόντα καταναλωτών είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαστε υπέρ της σημερινής πρότασης για το CMU. Τώρα όσον αφορά τους ε, συνταξιούχους και τα καλύτερα κέρδη. Εδώ θα έπρεπε να καθοριστεί η κατάσταση. Και όσο οι κεντρικές τράπεζες δεν αυξάνουν τα επιτόκια, οι συνταξιούχοι και άλλοι αποταμιευτές θα είναι χαμένη. Είναι αυτό που είπα και πριν. Είμαστε στη χειρότερη δυνατόν κατάσταση οικονομικά. Καταστολής δηλαδή, οικονομικής καταστολής. Δεν συμφωνούμε απόλυτα με την διάγνωση όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση για το CMU. Αυτό που προσπάθησα να πω και νωρίτερα είναι ότι Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη, χρειάζεται καταναλωτέ να ανοίξουν το πορτοφόλι τους, κάτι που δεν κάνουν πια. Και να έχουμε υπόψη μας ότι η κατανάλωση είναι τα δύο τρίτα του ΕΠ. Είναι δηλαδή η κινητήρια δύναμη πιο σημαντική που χρειαζόμαστε για να μπούμε και πάλι σε κανονική ροή. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Ναι, συμφωνούμε και εμείς για τη μόκλευση. Είναι όντως ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτώ και το ρολόι διότι είναι περασμένες 4.30. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές ε, που ήρθαν και μας μίλησαν για τις προκλήσεις στην ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς. Ακούσαμε λοιπόν ε, από ε, τράπεζες ασφαλιστικές εταιρείες από μία μη κυβερνητική οργάνωση της απόψεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέλφους που ήταν σήμερα παρόντες, που συμμετείχαν τόσο ενεργά στο, στη συζήτηση. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε γενική απελευθέρωση. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερη διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος των κινδύνων και το είδος των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε θα πρέπει να επικεντρωθούμε μάλλον περισσότερο στους γενικούς στόχους μας, στις γενικές αρχές μας και από τους σημερινούς ομιλητές ακούσαμε ποια είναι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή και τι δυνατότητες βελτίωσης υπάρχουν. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή ακρόαση. Τελικά, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πάζελ διαφορετικών ρυθμίσεων, όπως έχουμε βέβαια και αυτή τη στιγμή, αλλά το παζλ αυτό να δίνει μια συνολική εικόνα. Ο συζητητής ε, θα συνεργαστώ και με τους σκιώδεις συζητητές ε, τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες και ελπίζω τελικά να έχουμε μια καλή έκθεση πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας για τις ε, παρουσιάσεις σας. Και περνάμε τώρα στην, ε, στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης και μετά θα έχουμε ανταλλαγή, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, σχετικά με την έκθεση αυτή. Διακοπή ενός λεπτού. Dear colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Πρέπει να αρχίσουμε. Οι εμπειρογνώμονες μας, το προηγούμενο πάνελ φεύγει, αποχωρεί. Περνάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Δημόσια ακρόαση για το Target 2, Securities. Τίτλοι. Καλωσορίζω τον κύριο Ιβμέρς που είναι μέλος Εκκλησικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Δέχτηκε να μας μιλήσει για το Target 2 Securities. Πρόκειται για την πλατφόρμα διακανονισμού που αναπτύσσεται από το ευρωσύστημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τάπεζα συμμετέχει. Η ΕΚΟΝ λοιπόν σας προσκάλεσε 22 Ιουνίου έχουμε το πρώτο στάδιο μεταφοράς από τη χώρα μου την Ιταλία αλλά και σε διάφορες άλλες χώρες. Θα λάβει χώρα αυτή η αλλαγή και στη συνέχεια η Η μετάπτωση αυτή λοιπόν θα λάβει χώρα και θα αλλάξει η κατάσταση. Έτσι αν τα διάφοροι φραγμοί που υπάρχουν στην αγορά πρέπει να αναρμονιστούν οι πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και θέλουμε να ενισχύσουμε και την οικονομική σταθερότητα. Θα σας ακούσουμε λοιπόν όσον αφορά την εναρμόνιση των αγορών και βέβαια θα έχουμε και ερωτήσεις για το συνδυασμό με τον κανονισμό όσον αφορά τους τίτλους που εγκρίθηκε πέρυσι και επί το οποίο το Κοινοβούλιο ήταν ε, από κοινού υπεύθυνο. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε έτσι το ψήφισμα. Λοιπόν, κύριε Μέρς, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε καταρχήν να έρθω εδώ και να μιλήσω για το Target 2 Securities. Θυμάμαι πολύ καλά πόσο πολύ είχε υποστηρίξει το Κοινοβούλιο και παλιότερα την ιδέα αυτή. Πράγματι πήρε πολύ καιρό να εφαρμοστεί η αρχική αυτή ιδέα και να προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες. Τρεις μέρες μένουν μέχρι να πάρει σάρκα και οστά το σχέδιο αυτό. Την επόμενη Δευτέρα, πέντε εθνικά CSD θα περάσουν σε μετάπτωση βάσει των σχεδίων μας. Και βέβαια αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα, γιατί στο τέλος θα έχουμε 21 εθνικές πλατφόρμες που θα έχουν περάσει στην ενιαία. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Ευρωσυστήματος. Από την άλλη βέβαια, το πιο σημαντικό ήταν η εισαγωγή των backnotes και η δημιουργία και ο σχεδιασμός της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Μόντους operandi. Νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο σχέδιο, το SSM, που ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλο, αλλά η στιγμή ήταν πολύ συγκεκριμένη που πετύχαμε μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε αυτή τη νέα διάσταση ευρωπαϊκής συνεργασίας, ενιαίος επαπτικός μηχανισμός λοιπόν το SSM. Σήμερα έχουμε ένα σχέδιο ένα που είναι πιο κοντά είναι ο μηχανισμός αυτός του ευρωπαϊκού συστήματος, κάτι σαν τετραυλικά του. Το 1991 όταν αρχίσαμε με το ECP είχαμε εθνικά συστήματα. Και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε τότε είναι να συνδέσουμε τα διάφορα εθνικά συστήματα. Και αυτό ήταν που ονομαζόταν σύστημα Target. Αυτό το σύστημα Target ε, συνέδει τις πληρωμές των ε, διαφόρων εθνικών συστημάτων. Πολύ γρήγορα όμως είδαμε ότι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα είναι κάτι πολύ καλύτερο από ένα σύστημα διασύνδεσης εθνικών λύσεων. Συνεπώς, το 2004 είχαμε φτιάξει μετά το Target 1, το Target 2 και το Target 2 σε σχέση με το Target 1 ήταν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Όμως, πρόκειται για 56.000 τράπεζες που συνδέονται παγκοσμίως επιπλέον με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 2014 90 εκατομμύρια πληρωμές σε ρευστό και κανονίστηκαν στην πλατφόρμα αυτή με ένα τζίρο περίπου 503 ευρώ. Η χρήση του Target 2 είναι υποχρεωτική για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ιδιωτικές συναλλαγές. Θα έλεγα ότι είναι ακριβώς χάρη στις συμβουλές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το Target 2 σήμερα δεν είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται μόνο για το ευρώ, αλλά χρησιμοποιείται και για άλλα νομίσματα. Το Target 2 είναι για τους τίτλους και είναι κάτι που θα φροντίσουμε και στο μέλλον. ώστε και οι τίτλοι Target 2 να έρθουν πιο κοντά. Αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή υποδομή για πληρωμές σε ρευστό είδαμε ότι στο χώρο του ευρώ όλες οι πληρωμές γίνονται και με γκίσεις, με collaterals. Και δεν έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τίτλους. Αν λοιπόν θέλετε μια πληρωμή που ήταν εγγύηση, είναι καλύτερα να έχουμε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα Συγχρόνως όμως η Εθνική Πλατφόρμα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό των ε, τίτλων. Κάτι το οποίο μας οδήγησε να σκεφτούμε μήπως έπρεπε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα για ρευστό και τίτλους συγχρόνως. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα των τίτλων Target 2. Η Ευρώπη όπως γνωρίζετε, έχει πολλά εθνικά συστήματα, πάνω από 30 CSD. Έχει διαφορετικά συστήματα διακανονισμών, διαφορετικούς νόμους που διέπουν ε, τους τίτλους και διαφορετικούς κανόνες για διαδικασίες post-rate. Το πλονέκτημα ενός ολοκληρωμένου συστήματος είναι προφανές περισσότερη ασφάλεια, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, γιατί διακανονίζονται σε ε, χρήματα κεντρικών τραπεζών οι τίτλοι. Θα επιτρέψει οικονομίες κλίμακας, χωρίς να υπάρχει απέτηση συγχώνευση σε εθνικό επίπεδο. Πάντα τα εθνικά CSD είναι τα σημεία εισόδου βάση του ορισμού CSDR. Τα εθνικά CSDs, λοιπόν, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, αποτελούν μια προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι ένα στοιχείο που πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε είναι την διακυβέρνηση που έχουμε σχεδιάσει προκειμένου να πετύχουμε αυτή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στους τίτλους. Αν είχα ένα διάγραμμα, θα λέγατε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο αλλά και η Ευρώπη δεν είναι περίπλοκη με τόσες διαφορετικές πραγματικότητες που έχει. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε μια δομή διακυβέρνησης με εκατοντάδες οργανισμούς που συμμετέχουν. Φυσικά και είναι περίπλοκο. Όμως τελικά ήταν κάτι πλήρες που λειτουργήσε και θα έλεγα ότι είναι και μία από τις προϋποθέσεις για να πετύχει το σχέδιο αυτό. Η δέσμευση όσων συμμετείχαν σε αυτό το πλαίσιο, θα το έλεγα συνεταιριστικό, είναι κάτι που αποτελεί και ακριβώς τη δύναμη του σχεδίου. Ίσως να έχετε ήδη ακούσει κάποιες διαδόσεις ότι η πλατφόρμα T2S δεν ήταν αρκετά σταθερή. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η πλατφόρμα δηλώθηκε σταθερή και έτοιμη να αποκτήσει σάρκα και οστά και αυτό το είπε και το Συμβουλίο της και η ηγεσία της και τα CSD στα steering bodies. Αντιλαμβανόμαστε ότι το T2S θα έχει επιπτώσεις στις οικονομικές αγορές, χρηματοπιστωτικές αγορές και μετά από το C πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει απρόσκοπα. Αφού αξιολογήσουμε την πλατφόρμα όσον αφορά τη σταθερότητά της και το κατά πόσο είναι έτοιμη να της δώσουμε πνοή, θα είναι έτοιμη και για την μετάπτωση και αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και είναι κάτι που έχει επιβεβαιωθεί μετά από τις τελευταίες αξιολογήσεις που έχουν γίνει και που τις πήραμε σήμερα το πρωί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που θα υποβληθούν αύριο και στο Συμβούλιο δικητών. Βέβαια αυτό δεν αρκεί για να είναι έτοιμο το ευρωσύστημα. Χρειαζόμαστε και το εθνικό επίπεδο να είναι έτοιμο, που αποτελείται από τα CSD και από τις τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με το CSD. Αυτό που είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα είναι ότι πέντε χώρες έχουν οριστεί να συμμετέχουν στο πρώτο κύμα σε θελοντική βάση, που είναι η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Ελβετία και η Ιταλία. Όλα τα κεντρικά αποθετήρια των χωρών αυτών έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι έτοιμα και ότι θα αρχίσουν να κατεβάζουν όλα τα στατικά δεδομένα. Ό,τι δηλαδή συμβεί σε αυτές τις χώρες θα φορτωθεί σε μία νέα πλατφόρμα. Σε τέσσερις χώρες ο διακανονισμός των ε, συναλλαγών που θα έχει πάει σε αυτή την πλατφόρμα θα αρχίσει να είναι διαθέσιμο την Κυριακή. Οι Εθνικέ κοινότητε τραπεζών είπαν ότι θέλουν περισσότερο χρόνο για να δοκιμάσουν το περιβάλλον και γι' αυτό ζήτησαν η πλατφόρμα να αρχίσει από τη Δευτέρα, αλλά τον τελικό διακανονισμό όλων των trading, όλων των συναλλαγών να γίνει αργότερα, στα τέλη του Αυγούστου. 31 Αυγούστου φέτος. Η λύση αυτή έγινε αποδεκτή και από τους υπόλοιπους, γιατί μπορείτε να φανταστείτε αμέσω ότι αν υπάρχει μια καθυστέρηση στο πρώτο κύμα, αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει και το δεύτερο κύμα. Εμεί πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα είναι σταθερή, τουλάχιστον έτσι πιστεύουν τα κεντρικά αποθετήρια, οι συμμετέχοντες, ότι δεν θα επηρεαστεί το δεύτερο κύμα και αν υπάρχει μια ομάδα εργασίας η οποία θα αναφέρει μέχρι τους επόμενους μήνες, έτσι θα δούμε αν πρέπει να αντιμετωπιστεί και κάποιο άλλο πρόβλημα. Ομόφωνα υπήρχε απόφαση οι Ιταλικές τράπεζες να έχουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου πριν ε, φορτώσουν παντελώς τα στοιχεία τους σε αυτή την κοινή πλατφόρμα. Τώρα, Πλέον ακτήματα παρουσιάζει τώρα αυτή η ενιαία πλατφόρμα. Όπως τα εθνικά αποθετήρια θα οδηγήσει την ατζέντα το θεματολόγιο της εναρμόνισης. Έχουμε ακόμα υπερβολικό κατακαιρματισμό των εθνικών αγορών στην Ευρώπη και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε εναρμόνιση και ίσως και πλήρη εναρμόνιση είναι μια διαδικασία που οδηγείται από την αγορά που θα επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε όλο το δυναμικό της αγοράς τίτλων. Το 2001-2003 νομίζω θυμόσαστε την έκθεση Τζοβαϊνή που τόνιζε όλες τις δυσκολίες που είχαμε για, για το διακανονισμό μετά από μια συναλλαγή τίτλων και από αυτά τα προβλήματα που ανέφερε η έκθεση Τζοβανίνη το T2S και τα αποθετήρια τίτλων θα αντιμετωπίσουν πολλά από αυτά τα προβλήματα. Παραμένουν όμω ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί και ελπίζουμε ότι η συζήτηση για την Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει εν καιρό και, και είμαι έτοιμο να συζητήσω μαζί σας τι πρέπει να κάνουμε και ποια είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και είμαι έτοιμος για τα ερωτήματα που τυχόν θα είχατε. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρόεδρος, κύριε Μέρσια, για την παρουσίασή σας και ξεκινάμε τώρα με τις ερωτήσεις και με τον κύριο Μπέρντ Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέρσ. Νομίζω ότι έχετε ένα πολύ σημαντικό έργο μπροστά σας Ήδη το 2008 ξεκίνησε η απόφαση για τη δημιουργία αυτού του εργαλείου. Μετά από 7 χρόνια, όπως είπατε, μπορείτε να ξεκινήσετε με 4,5 κράτη-μέλη, γιατί η Ιταλία μέχρι το καλοκαίρι δεν θα συμμετέχει ακόμα στο σύστημα αυτό και πρέπει να περιμένετε λιγάκι για να την ενσωματώσετε πλήρως. Εγώ, εγώ φυσικά, μεγάλη εκτίμηση για αυτό το τεράστιο οργανωτικό έργο που έχετε κάνει και μετά από αυτά τα οποία είπατε ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Ποια ήταν η αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα και βλέπουμε στον κατάλογο ότι μέχρι το 2017 θα έχουμε τρία μη κράτη της ζώνης του ευρώ, Δανία, Ουγγαρία, ακόμα και την Ελβετία. Πώ βλέπετε τώρα εσεί τη δυνατότητα, αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα, Χώρε όπω η Μεγάλη Βρετανία παραδείγματο χάρη που έχει μεγάλη σημασία στον χρηματοπιστωτικό χώρο να συμμετάσχει ή εκεί πέρα υπάρχει ανταγωνισμό με την πλατφόρμα σα. Μπορεί τώρα να συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να υπάρξει σύγκληση μεταξύ των πλατφορμών αυτών και να υπάρξει κάποια θετική συνεργασία στο μέλλον. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σα θέσω. Το σύστημα Target είχε αντιμετωπίσει μεγάλες αντιπαραθέσεις σε σχέση με τους ε, ενδεχόμενους κινδύνους. Υπήρξαν επιστημονικές λοιπόν αντιπαραθέσεις, έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θυμόσαστε ότι ο καθηγητής Ζιν από το, μόναχο, το ύφο του μονάχου είχε διατυπώσει πολλές κριτικές για το σύστημα για το Target 2 και εσείς μιλάτε τώρα για ένα όγκο συνολικό 500 δισεκατομμύριων ευρώ. Είναι τόσο μεγάλος λοιπόν ο όγκος των συναλλαγών που θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχετε και μια πλατφόρμα που λειτουργεί σε πολλά νομίσματα και όχι μονάχα σε ευρώ. Πώς βλέπετε λοιπόν το μέλλον αν προχωρήσουν όλα βάσει του σχεδίου. Μέχρι το 2017 μπορούμε να έχουμε και περισσότερο όγκο συναλλαγών και μπορεί να είναι και ένα παράδειγμα όπως το αντίστοιχο αμερικανικό σύστημα και πώς προχωρούν και οι συζητήσεις για την πλήρη κατάργηση των χαρτονομισμάτων και κερμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα θυμάστε ότι στην αρχή είχαμε σκεφτεί ότι δεν μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε την αγορά να, ε, πάρουν, να πάρει μέτρα για τέτοια πλατφόρμα ως ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά μετά από παρατήρηση κάποιων ετών και αφού διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν δυσκολίες να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια σε σχέση κυρίως ε, με το ρυθμιστικό περιβάλλον του δημοσίου τομέα αποφασίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να ε, προχωρήσει στη δημιουργία μια τέτοια ε, πλατφόρμα και μάλιστα ε, ήταν αυτή λόγω της συναλλαγματικής πολιτικής, της νομισματικής συγγνώμη πολιτικής ήταν ακριβώς ο θεσμός ο οποίος περισσότερο εξαρτάται από, την, από τις αποτελεσματικές δομές πληρωμών πριν από 15-10 χρόνια συμπεράναμε εν τέλει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Γενική Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει και να πάρει τις αποφάσεις ε, βεβαίως. Θα πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο και να του απονείμουμε τα εύσημα για την συμβολή του, γιατί το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως α, επέμεινε ότι θα έπρεπε να είναι πλατφόρμα όχι μόνο για το ευρώ, αλλά για πολλά νομίσματα. Στην αρχή βεβαίως αυτό οδήγησε σε κάποιες λειτουργικές επιχειρησιακές ε, ε, δυσκολίες και περιπλοκές, αλλά εν τέλει ε, έγινε και πιο ελκυστική πλατφόρμα. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από δύο-τρεις εβδομάδες επισκέφθηκα την ε, Κεντρική Τράπεζα της ε, Σουηδίας ε, γιατί είναι κεντρική τράπεζα η οποία είναι υπεύθυνη για το κεντρικό νόμισμα και για την συμμετοχή του νομίσματος σε αυτή την πλατφόρμα αλλά είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη και για την, ε, ε, για την απόθεση τίτλων σε μερικές περιπτώσεις, σε ορισμένες χώρες δηλαδή, ε, δεν εξαρτάται το αποθετήριο τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αναθεωρούν λίγο την άποψή του σχετικά με την συμμετοχή στο TTS και είναι μια θετική εξέλιξη. Αυτό είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο. Βεβαίως δεν μπορώ να σας κρύψω ότι αυτό ε, κινήθηκε κιόλας από το γεγονός ότι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της ε, Σουηδίας παρακολουθεί στενά τις τεχνικές εξελίξεις σε άλλες ε, χώρες, άτακτες χώρες όπως η Φιλανδία. Και ε, και ε, εάν ε, το φιλανδικό σύστημα γίνει συμβατό με το Target 2, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει και η Σουηδία οι συνάδελφοι της Κεντρικής Τράπεζας από την ε, Νορβηγία επίσης ε, θα ξαναδούν φαντάζομαι την, την απόφαση τους ε, σύντομα γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί θα πρέπει να στραφούν προς το target του security λόγω του περιβάλλοντος το οποίο θα κινούνται όσον αφορά ε, ε, το θέμα αυτό μπορώ να πω ότι έχουμε άλλους δύο συμμετέχοντες που θα ε, έρθουν μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου για την location policy και μετά από απόφαση και του Βρετανικού δικαστηρίου διότι βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ενδιαφέρον ε, να ε, δουν την δυνατότητα χρήσης του Target 2, κυρίως για τα CCPs που ήδη λειτουργούν σε ευρώ, αλλά που βρίσκονται στο Λονδίνο. Θα πρέπει να δούμε εάν ε, θα καταλήξουμε κάπου αλλά ήδη έχουμε αποφασίσει να ενδυναμώσουμε την ε, συνεργασία μας όσον αφορά τέτοιου είδους υποδομές της αγοράς και βεβαίως ε, αυτή, αυτό είναι και το πλεονέκτημα των ε, ολοκληρωμένων ε, ε, υποδομών γιατί με τον τρόπο αυτό ε, μπορούν να υπερκεραστούν διάφορα προβλήματα και να έρθουμε σε επαφή με τις εθνικές αρχές. Επίσης μας ρωτάτε εάν ο στόχος 2 θα κινηθεί προς διαφορετικά νομίσματα. Ξεκινήσαμε με το Target του security γιατί αυτό το σκέλος έχει το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκτός Ευρώπης. Ε, είτε σε ευρώ είτε σε, ε, στο δικό τους νόμισμα. Μπορούν να το κάνουν ε, χρησιμοποιώντας το δικό τους κεντρικό αποθετήριο τίτλων στα πελέσια του TTS είτε είτε είτε Uh, ε, είτε χρησιμοποιώντας ε, το, ε, την ρευστότητα έτσι, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα υφιστάμενα ε, προβλήματα ε, και μετά να υπάρχει μετάπτωση των άλλων ε, σημείων των Ευρωπαίων συμμετεχόντων αλλά βεβαίως κάθε φορά θα πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το συμφέρον ή το ενδιαφέρον που θα έχουν μη ευρωπαϊκά κεντρικά αποθετήρια να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ να υπενθυμίσουμε ότι επειδή είναι πολλές οι ερωτήσεις, ε, πέντε λεπτά ο καθένας, ο κύριος Τάγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα αυτό. Αξίζει τον κόπο όμως να ασχοληθούμε με αυτό. Στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, λίγο πριν την έναρξη λειτουργία του συστήματος, σκέφτεται κανεί τι θα μπορούσε να πάει στραβά. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχετε εξετάσει τους κινδύνους. Αλλά από την άλλη θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θέλετε ένα σταθερό περιβάλλον ε, και δεν θέλετε κι εσείς να διακινδυνεύσετε να έχουμε μια πλατφόρμα που να μην λειτουργεί. Καταλαβαίνω τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Αλλά πώς έγινε η επιλογή. των ε, χωρών ε, ε, εθελοντικά συμμετείχαν και επίσης βλέπω ότι υπάρχει και ελληνική συμμετοχή. Η ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ε, ε, είναι μάλλον ένα τρικυμιώδες περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει λοιπόν με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας. Και τέλος θα μπορούσατε παρακαλώ να αναπτύξετε αυτό που είπατε σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν εντός της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, δεν πιστεύουμε ότι θα πάει τίποτα στραβά. Σε ένα πρόγραμμα τέτοιου τύπου είναι προφανές ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρχουν κάποια προβληματάκια κατά τις δοκιμές. Σταματήσαμε την προσαρμογή του λογισμικού πριν δύο εβδομάδες, διότι είχαμε ακόμα και τότε κάποια προβληματάκια, τα οποία όμως δεν θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Για καθένα από αυτά τα προβληματάκια είχαμε λύση. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εμείς αλλά και οι χρήστες Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην έναρξη λειτουργία του συστήματος. Κατά τις... το πρώτο διάστημα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα διάφορα προβληματάκια ώστε να ε, λειτουργεί επιτυχώς κατά 100% και όχι κατά 99,8%. Ε, δεύτερον, ε, όπως είπα, ε, εθελοντικά αποφασίστηκε ποιος θα συμμετάσχει με συζήτηση μεταξύ των διαφόρων συμμετοχόντων. Δεν ε, ε, επιβλήθηκε σε καμία χώρα να συμμετέχει στην πρώτη ή στη φάση. Αυτό αποφασίστηκε στο συνεργατικό κλίμα που ε, επικρατεί. Τρίτον, όσον αφορά την Ελλάδα, και το BOGS. Ε, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλλει στην ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι αγαθό το οποίο χρειάζεται όλη η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα. Η συμμετοχή λοιπόν της Τράπεζας της Ελλάδας συμβάλλει στην σταθεροποίηση στην Ελλάδα και μεταξύ Ελλήνων συμμετεχόντων αλλά και μεταξύ Ελλήνων και μη Ελλήνων ε, εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Για να λειτουργούν τα πράγματα ομαλά. Νομίζω δηλαδή ότι είναι προς όφελος όλων. Τέλος, σε τι βαθμό αυτό συμβάλλει στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Καταρχάς αντιμετωπίζονται έτσι κάποια από τα τελευταία εμπόδια της έκθεσης Τζοβανίνη για την ευελτιστοποίηση των αγορών μας. Γιατί έτσι έχουμε εναρμόνιση, έχουμε καθορισμό ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων και ακόμα στην Ευρώπη έχουμε υπερβολικά μεγάλο κατακαιρματισμός της υπηρεσίας ολοκλήρωσης των συναλλαγών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν στην εξάλληψη αυτών των διασυνοριακών εμποδίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε την Κέις Βίνπεν που είναι η συγγήτρια για τον κανονισμό του για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μέρς. Ε, ε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ε, ε, νιώθω μεγάλη χαρά που επιτέλους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αυτό. Έχω περάσει πολλά χρόνια ασχολούμενη με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι εσείς έχετε δαπανίσει ακόμα περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να θέσετε σε λειτουργία το πρόγραμμα αυτό. θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ που μπορείτε τώρα σύντομα να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα. Αυτό δείχνει ακριβώς ε, πόσο αποδίδει η επιμονή και η για τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα λειτουργήσει σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα αυτή θα έχει τη δυνατότητα να διευρυνθεί. Ως εισηγήτρια όμως ε, για τον κανονισμό για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ε, δεν μπορώ παρά να ζητήσω τη συμβουλή σας για ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει ο κανονισμός ε, αυτός έχει εμπνευστεί σε μεγάλο βαθμό από τα target του securities ε, και προσπαθούμε να έχουμε ένα βιβλίο κανόνων για το σύνολο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρότυπα, τα πρωτόκολλα και θέλουμε έτσι να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τα ωφέλη από το target ε, του Security. Ωστόσο, κάποιοι κανόνες εντός του κανονισμού για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων που θέλαμε να συνδέσουμε με την εφαρμογή του target του Security... ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τον διακανονισμό τίτλο, ε, μας φέρνει αντιμέτωπους σε ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος. Τι γίνεται σε περίπτωση αποτυχίας του διακανονισμού. Πιστεύω ότι μπορεί οι πράξεις να διεξάγονται πολύ πιο ομαλά εάν ε, το CSTR, ο κανονισμός αυτός, ε, συνδεθεί με την τελευταία φάση λειτουργίας ε, και εφαρμογής του target του securities, ώστε να αποφύγουμε και την επικάλυψη δαπανών. Η ερώτηση μας λοιπόν είναι, συμφωνείτε με την καθυστέρηση αυτή θα συμφωνήσετε με την αναβολή αυτή και δεύτερον θα πρέπει να αναφερθώ και στην ερώτηση του συναδέρφου Βενελάνγκε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός τρόπος να μειώσουμε το κόστος του διακανονισμού για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο θα ε, φέρει ωφέλη σε όλα τα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα αυτό είναι θελοντικό, δεν ε, αναγκάσαμε κανένα να συμμετάσχει και γι' αυτό ε, δεν ένιωσε κανείς την ανάγκη να προστατεύσει το εθνικό του σύστημα. Πόσο καιρο, πόσος καιρός νομίζετε ότι θα χρειαστεί για το δικό μου κράτος μέλος και για τα άλλα να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή για τους διακανονισμούς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και για τη στήριξή σας. Οι ενιαίοι κανόνες διακανονισμού είναι αυτό που θέλουμε, γιατί έτσι είναι κοινή στόχη μας με το CSDR. Υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου είμαστε συμπληρωματικοί με το CSDR για πιο ολοκληρωμένα συστήματα, πλατφόρμες. Όσον αφορά το κατά πόσο πρέπει να καθυστερήσουμε την εφαρμογή μέχρι το τελευταίο κύμα, ε, προφανώς θα βοηθήσει να αποφύγουμε να έχουμε ένα διπλό καθεστώς για αυτούς που δεν έχουν ακόμα κάνει μετάπτωση με αυτούς που έχουν κάνει τη μετάπτωση. Από την άλλη βέβαια η εμπειρία μου με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ότι πάντα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε την ε, πειθαρχία στην προθεσμία και να την καθυστερήσουμε. Αν υπάρχει πίεση που διατηρείται προκειμένου η εφαρμογή να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα χωρίς να υπάρχει σύστημα κυρώσεων για αυτούς που δεν είναι έτοιμοι, ε, θα πετύχουμε έτσι το ίδιο αποτέλεσμα. Πάντως, θα ήθελα να είμαι σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στον τομέα αυτό έχει αποδειχτεί μια μεγάλη στήριξη και τέρος μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάπτωση του T2C. Οι συζητήσεις βέβαια θα συνεχιστούν. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπα, Είμαστε σε καλές επαφές με την Τράπεζα της Αγγλίας προκειμένου να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικότητα, σε υποδομές, σε συνεργασία, εποπτεία, προκειμένου ο ευρωπαϊκός χώρος να είναι περισσότερο ασφαλής, περισσότερο αποτελεσματικός και να στοιχίζει και λιγότερο στους παίκτες της αγοράς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. ο δεμάς, είναι ο επόμενος ομιλητής. Δεν βλέπω κανένα από τους φιλελεύθερους, ναι. Είναι κάπως ε, το αποτέλεσμα της έκπληξης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, λοιπόν. ήθελα να εστιάσω σε μια διαφορετική πτυχή του Target 2. Ο Βέρνε Λάγκερ μίλησε ήδη για το Hans-Werner Zinn. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τους κινδύνους του τι θα συνέβαινε αν ένα κράτος μέλος χρέοκοπούσε ή έπαβε να ε, ξεπληρώνει τα, τα οφειλόμενα ποσά στο Target 2. Είναι φυσικά και όπως είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ότι έχουν υπάρξει σημαντικές ροές και φυγές κεφαλαίου που φυσικά οδηγούν και σε, σε τόκο που πρέπει να καταβληθεί στα καθυστερούμενα ποσά που πρέπει να αποκληρώσει μια χώρα. Θα ήθελα όμως να ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο κούρεμα ή κάτι άλλο σε σε σχέση με αυτά τα υπο, υπολοιπόμενα ποσά και οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι με το σενιοράζ, με, με τα έσοδα από την ε, έκδοση ε, νομίσματος μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν. I... Ναι, λέει ο κύριος ε, Μέρς. Εγώ θα πρέπει να διαφωνήσω λιγάκι. Το Target 2 δεν αντανακλά μονάχα κεφαλαίωκες κινήσεις. Αυτό συμβαίνει μονάχα αν μια χώρα έχει χάσει απολύτως την πρόσβαση στις ε, κεφαλαιακές αγορές. Κάτι το οποίο κοντεύει να γίνει πραγματικότητα για μια χώρα, αλλά μια χώρα που έχει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, το ΤΑΦ 2 σίγμα εκφράζει μονάχα ένα τμήμα της πρόσβασης ε, στις αγορές και υπάρχουν οι διατραπεζικές ροές οι οποίες ε, δεν θα βέβαια ε, εμφανίζονται πλήρως στην, ε, στον ισολογισμό των κεντρικών τραπεζών. Αλλά οι τράπεζες μπορούν να κάνουν και δανειοδοτήσεις διμερού, διμερούς επίπεδου διατραπεζικές. Το πολιτικό τμήμα του ερωτήματος όμως τώρα είναι τι θα συμβεί αν μια χώρα βγει από τη ζώνη του ευρώ. Εγώ λέω ότι αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη και εμεί θεωρούμε ότι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ είναι αμετάκλητη και βασιζόμαστε σε αυτήν την ιδέα. Έτσι έχει διατυπωθεί η συνθήκη και έτσι έχουν διατυπωθεί και οι κανονισμοί μας. Αν τώρα θελήσουμε να εισαγάγουμε ένα σύστημα που κατά την άποψή μας θα οδηγούσε σε επανεθνικοποίηση και τότε θα θέταμε να αμφιβόλο το αμεκτάκλητο του ευρώ, τη συμμετοχή στο ευρώ. Βέβαια υπάρχουν και μηχανισμοί όπως αυτός ο οποίος υπήρχε στις ΗΠΑ που δεν είναι ένας πλήρης μηχανισμός για τον διακανονισμό των υπολείπων στο τέλος του χρόνου αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες ε, δια, διατάξεις για να μπορέσει να διατηρηθεί κάποια μεγαλύτερη ε, προληπτική εποπτεία για τα ε, υπολείμματα για τα οφειλόμενα ποσά από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά από το σχεδιασμό το αναρχικό του συστήματος τα οφειλόμενα ποσά του Target 2 δεν παραμένουν εκρεμή χωρίς διακανονισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν τώρα κάποια κάτι μέλη παραμένουν διαρθωτικά με ελληματικό ισοζύγιο στο Target 2 και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ευθυγραμμίζεται με την ιδέα ενός ευρωπαϊκού συστήματος, ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος όπου πρέπει να υπάρχει και μια σύγκληση, μια πραγματική σύγκληση μέσω της ευθύνη της κάθε χώρας. Όσο έχουμε λοιπόν αυτή την αρχή της ίδιας ευθύνη, άγγενα Antwortung, την οικονομική δραστηριότητα, τότε, μάλλον, τότε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα της διακυβέρνησης και τότε δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουμε το σύστημα των ε, ισοζυγίων του Target 2. Αλλά μπορεί να παραμείνει όπως έχει τώρα. Αν περάσουμε σε ένα σύστημα όπου θα υπάρξει ένας επανακαθορισμός του συστήματος, αυτό μπορεί να είναι πιο αποσταθεροποιητικό παρά η παραμονή στο τρέχον σύστημα. Και για τη δήλωσή σας ότι ένα, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να έχει αρνητικό κεφάλαιο, υπήρξανε και τέτοια παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το γεγονός καθεαυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα έχει άμεσες χρηματοπιστωτικές συνέπειες μεν, αλλά θα μπορούσε να υποσκάψει την φήμη μιας κεντρικής τράπεζας στα μάτια του κοινού. Και επομένως μια κατάσταση αρνητικού κεφαλαίου μπορεί να είναι προσωρινά δυνητικά ε, εφικτή αν εξηγηθεί καλά στους καταναλωτές και συνάδει με την κατάσταση μιας χώρας οικονομικά, αλλά δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να σας συγχαρώ για την ε, δημιουργία αυτής της νέας υποδομής με τόσο γοργό ρυθμό. Ε, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος εργασίας που απαιτήθηκε. Η ερώτησή μου για το target του security είναι αν σε γενικές γραμμές ε, κατά την άποψή σας ε, ένα σύστημα target του ε, security χωρίς το ευρωπαϊκό, χωρίς το Βασίλειο στην Ένωση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και να είναι αποτελεσματική. Όσον αφορά το Target 2, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνάδελφος Ντεμάζη ήδη υπέβαλε το ερώτημα, θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα. Εσείς απαντήσατε μάλλον με πολιτικό τρόπο ε, και το light motif το ακούσαμε ότι το ευρώ δεν διαλύεται και τα λοιπά και είναι αμετάκλητο. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς ε, να μην σκεφτεί ότι έστω και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες θα μπορούσε να προκύψει η περίπτωση μιας χώρας η οποία μονομερός αποφασίζει να εγκαταλείψει το ενιαίο νόμισμα. Και αν μιλήσουμε ε, έξω από τα δόντια, η περίπτωση της Ελλάδος ας πούμε είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα μπορούσε, ε, μάλλον το ενδεχόμενο να βγει η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τι θα γίνει τώρα τότε λοιπόν με το Target 2 ε, το οποίο ήδη έχει ένα αρνητικό 99 δις ευρώ. Οι τράπεζες των άλλων κρατών που παραμένουν μέρη της Ευρωζώνης και της πλατφόρμας θα έχαναν χρήματα ή θα ήταν στην ουσία μια θεωρητική απώλεια η οποία απλώς θεωρητικά θα έμενε στους, θα φαινόταν στους προϋπολογισμούς. Επίσης, σε περίπτωση που η Ελλάδα μείνει έξω από το σύστημα Target 2, όχι με δική της απόφαση, θα μπορούσε να υπάρχει παραβίαση του άρθρου 63 όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση που εξωθηθεί εκτός ευρώ η ε, Ελλάδα ε, μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι ακόμα και αν δεν προβλέπετε τίποτα στη συνθήκη, δεν είμαστε προστατευμένοι κατά τις μονομερούς δράσεις. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα εθνικά προβλήματα. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι μια προσέγγιση συνεργασίας. Για να πετυχαίνουμε συμφωνία ακόμα και για δύσκολες καταστάσεις. Τα νούμερα που αναφέρατε είναι σωστά. Δεν θα ήθελα να κάνω υποθέσεις σχετικά με μια τέτοια κατάσταση. Δεν αποτελεί λοιπόν μέρος της υπόθεσής μας, αλλά εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ύπαρξη της Ευρωζώνης όπως αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο. Το να αρχίσουμε τώρα να κάνουμε υποθέσεις ότι το πολιτικό επίπεδο θα αλλάξει προσέγγιση, θα ήταν το λιγότερο μη σοφό από πλευράς ε, ενός τεχνικού εμπειρογνώμονα, ε, ενός θεσμικού οργάνου. Από τεχνικής άποψης όμως, αυτό θα σήμαινε ότι θα είχαμε χρέος μιας κεντρικής τράπεζας, το οποίο θα περνούσε στο λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το χρέος, το πώς θα αποπληρωθεί, θα αποτελεί αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Δεν προβλέπεται τίποτα όμως σχετικό αυτή τη στιγμή και σίγουρα όπως σας είπα, δεν περιλαμβάνεται στους προβληματισμούς μας και στις εργασίες μας. Η προσέγγιση μας προβλέπει διατήρηση της ε, συνδεκτικότητας ε, της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτά που μας είπατε δείχνουν ότι είναι προς συμφέρον όλων να αποφύγουμε συνέπειες πολύπλοκες για όλους και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύουμε ότι και αυτός είναι ένας ρόλος να συνεχίσουμε με αφοσίωση της εργασίας μας. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη η διευκρίνηση σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Ε, συμφωνούμε λοιπόν με την ακεραιότητα της Ευρωζώνης, όπως είπατε και εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την σημαντική συνάντηση, για τη συζήτηση. Όπως είπατε, το Κοινοβούλιο είναι θερμός υποστηρικτής ε, του προγράμματος Target to Securities. Θα παρακολουθήσουμε στενά τις ε, περαιτέρω εξελίξεις και αποτελεί το πρόγραμμα αυτό ένα πολύ καλό σημάδι, κάτι που σίγουρα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ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 Περνάμε στο σημείο 15 της σημερινής διάταξης. Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε Αντίκτυπος και μελλοντική πορεία προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα και προς μια ένωση των κεφαλαίων Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κρόαση τώρα. Περνάμε στη συζήτηση ανταλλαγή απόψεων. Το λόγο έχει ο συγητής. Μπούθαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν πολύ θετικό σήμερα το απόγευμα να ήταν πολύ καλό που είχαμε καταρχήν την ακρόαση και μετά τα, τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με εκπροσώπους του τραπεζικού και του ε, ασφαλιστικού τομέα της Finance Watch και από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Αυτό μας δίνει μια λοιπόν μια ε, μας δίνει την εντύπωση ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία πάνω στον κόσμο της ρύθμισης και της ανάγκης να έχουμε μια σφαιρική εικόνα και να δούμε αν κάποια στοιχεία θα πρέπει να αρθούν από αυτό το πλαίσιο. Η κρίση έδειξε τα κενά που υπήρχαν και τις ελλείψεις και υπάρχουν όλα αυτά τα παραθυράκια τα οποία πρέπει να τα κλείσουμε αργά ή γρήγορα. Η επισκόπηση αυτή λοιπόν δεν μας οδηγεί προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης απορρίθμισης, αλλά μια, μιας πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής ρύθμισης. Και γι' αυτό πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα την ε, τις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών για να δούμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νομοθετικές πράξεις που αυτή τη στιγμή είναι εν Έχουμε ψηφίσει πολλά νομοθετήματα για τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές με μια πρωτοφανή, αν θέλετε, πολυπικιλία ρύθμιση προϊόντων, Ινστιτούτων, αγορών και τα λοιπά, κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ρυθμιστών και εποπτικών αρχών. Ο στόχος όλης αυτής της ρύθμισης είναι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή προστασία στον καταναλωτή και όχι να τροποποιήσουμε την οικονομική, μακροοικονομική ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε την ρύθμιση και την νομοθετική αυτή ρύθμιση για το αν πράγματι πέραν του επιδιωκομένου στόχου έχει αρνητικά αποτελέσματα στην οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι μειώνεται η κερδοφορία του και όταν ένα μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών εταιριών αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολεύεται να ε, δεχτεί την έννοια μιας ευρωπαϊκής κεφαλαιοχικής αγοράς. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι μια συνολική αντιμετώπιση των νομοθετικών μέτρων θα πρέπει να γίνει. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε μια μελέτη, να ζητήσουμε μια μελέτη επιπτώσεων που να εξειδικεύει τους διάφορους τομείς, τον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό παραγωγός χάρη, αλλά τελικά θα πρέπει να καταλήξει και σε συμπεράσματα τα οποία υπερβαίνουν μια στενή τομεακή αντιμετώπιση και το είδαμε και αυτό από αυτά που μας είπαν οι πανελίστες μας. Πέρα λοιπόν αυτών κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και την πρακτική που έχουμε μέχρι τώρα για τις εκθέσεις αντικτύπου και να την επανεξετάσουμε τη μεθοδολογία αυτή. Η μεθοδολογία της Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες κατά τις οποίες βρίσκονται οι χρηματοπιστωτικοί φορείς και το μέγεθός τους. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι πολλές φορές οι εκθέσει αντικτύπου της Κομισιόν είναι μονάχα επιδερμικού χαρακτήρα. Συζητήσει για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε την ε, διαδικασία νομοθετικής ρύθμιση και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τα κενά και για να μπορούν όλα να λειτουργούν με κάποιο συγκροτημένο τρόπο μέσα στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Για μένα είναι απαραίτητη λοιπόν η συνεκτικότητα και η συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων και όχι η πολυπλοκότητα και η ασάφεια. Όλα αυτά φυσικά έχουν σημασία και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και επίσης μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πώς συνδέεται και συναρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις παγκόσμιες ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να μην έχουμε σημαντικές αποκλήσεις και επίσης είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και τη διαδικασία λήψης απόφασης και τις αρμοδιότητες το πώς παραδείγματος χάρη γίνεται η ρύθμιση σε επίπεδο τεχνικών προτύπων ή ε, εφαρμοστικών πράξεων. Επαναλαμβάνω βέβαια τον εαυτό μου όταν σας λέω ότι θα πρέπει από το παζλ που έχουμε με τους διαφορετικούς κανόνες και τις ρυθμίσεις θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο το οποίο βγάζει νόημα και σαν σύνολο και όχι μοναχά στις λεπτομέρειες τους. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους κοιόδης συζητητές στους επόμενους μήνες και πιστεύω ότι από τη βάση μιας καλής και γεμάτης εμπιστοσύνης συνεργασίας μπορούμε να καταλήξουμε και σε ένα θετικό αποτέλεσμα για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Φιλόδοξο πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό όμως. Ο πρώτος ομιλητής, ο κύριο Πολ Τάγκ, σκιώδης από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, ναι. Από φιλοδοξία, ναι. Και εγώ. Σήμερα μιλήσαμε για την ε, Κεφαλαϊκή Ένωση. Είναι μια προσπάθεια τα προβλήματα της κρίσης να τα ξαναδούμε υπό διαφορετική σημαία. Εξαρτάται βέβαια από την προσέγγιση μας απέναντι στην κεφαλακή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να είναι κατά ευκαιριών για πιο αποτελεσματικές αποταμιεύσεις, για μικρότερους κινδύνους, λιγότερους κινδύνους και να βελτιώσουμε την προοπτική της ανάπτυξης, της μακροχρόνιας ανάπτυξης. Είχαμε όμως χάος τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξυπηρετεί την οικονομία, κυρίως τώρα μετά την κρίση. Μετά λοιπόν τις πρώτες αισθήσεις που γίνονται για τον απολογισμό, θα έλεγα, το θέμα δεν είναι να πιστοχωρήσουν οι ρυθμίσεις, όχι. Είναι να κάνουμε έναν απολογισμό και να βρούμε τρόπους με τους οποίους να μπορούμε να βελτιώσουμε τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις προς όφελος, προς το συμφέρον των λόγων της Ευρώπης, που είναι και προς το συμφέρον του χρηματοπιστωτικού τομέα, γιατί έτσι θα εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Η έναρξη της συζήτησης είναι καλή Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Έτσι, έρχομαι σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το θέμα της συστημικής ισορροπίας το έχει εξετάσει κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά για να βελτιώσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι το έχουμε εξαντλήσει. Υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών. Εδώ ακόμα υπάρχει θέμα προκυκλικής αποσταθεροποίησης τέτοιων μηχανισμών. Άρα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση για την αστάθεια. Είναι ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. πρέπει να φροντίσουμε ότι υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση. Και ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα φαίνεται σαν ένα εμπόδιο, σαν κάτι κακό, αλλά σαν κάτι που διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα. Γιατί αλλιώ αν το πιστωτικό τομέα είναι ασταθή, έχει αποτύχει. Δεύτερον, είναι σημαντικό να δούμε και μια αλλαγή από τις οφειλές στην ανάληψη κινδύνου. Χρειαζόμαστε μια καινοτόμα οικονομία. Επιχειρήσεις που να είναι διατεθειμένες να αναλάβουν κινδύνους. Η αλλαγή προς τις κεφαλαϊκές αγορές είναι μια αλλαγή και προς την κατεύθυνση της ανάληψης κινδύνου και καινοτόμων επενδύσεων. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να κοιτάς μόνο την οικονομική ρύθμιση. Υπάρχει και το θέμα της φορολογίας που δίνει πλεονεκτήματα στις οφειλές, στη χρέωση δηλαδή, και αντίθετα μειονεκτήματα στην ανάληψη κινδύνου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η προστασία του καταναλωτή επίσης. Το άκουσα και από τον εισηγητή ότι η προστασία αυτή πρέπει να είναι στο κέντρο των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων. Παραμένουν ε, βέβαια πολλά να γίνουν για να βελτιωθεί αυτό. Πάντως συνάδει με το στόχο μας που λέει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να εξυπηρετεί τον κόσμο, την πραγματική αγορά, τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα είμαι σύντομο γιατί πολλές ιδέες βέβαια υπάρχουν για το τι μπορεί να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει. Όπως είπα, να έχουμε υπόψη μας τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, γιατί αν δεν είναι σταθερός θα έχει αποτύχει, όπως είπαμε, για την πραγματική οικονομία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πολ. Και Σούμπερτ, ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί συνδέονται εδώ τα δύο θέματα θέλουμε να κάνουμε απολογισμό των ε, χρηματοπιστωτικών κανονισμών που υλοποιήσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, το CMU δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η συνέχεια αυτών που κάνουμε και νομίζω ότι ε, ο κύριος Μέρσο, μάλιστα μας παρουσίασε το Target 2 Securities μια πλατφόρμα ε, ε, δηλαδή την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη η Ευρώπη. Και από τη στιγμή ε, και μάλιστα η ιδέα ότι οι αγορές είναι κάτι ε, ολοκληρωμένο μας πήρε 10 χρόνια να το καταλάβουμε ε, και ε, νομίζω ότι αυτός ο απολογισμός μαζί με τον μελλοντικό ECMU είναι μια πολύ καλή συζήτηση που πρέπει να γίνεται μαζί. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν και από το προηγούμενο πάνελ. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να δούμε τις ε, εξαιρέσεις που έχουμε βάλει στο επίπεδο 1. Ε, είχαν λόγο που μπήκαν αυτές οι εξαιρέσεις. Έπρεπε να μπουν έτσι ώστε να προστατευτούν κάποια άτομα. Βάλαμε επίσης εξαιρέσεις για τα συνταξιδετικά ταμεία, γιατί πραγματικά χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση και των ταμείων ταμείων και των χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων τους. Ε, Επίσης, ε, έχουμε κάποια ζητήματα όσον αφορά την συνέχεια και την συνεκτικότητα, ε, ε, γιατί υπάρχει μία διασπορά όσον αφορά τα νομοθετήματα στα οποία αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Είναι και στη ΜΥΦΙΤ, είναι και στην ΑΕΜΠΙΑΦ, είναι και γενικώ υπάρχει μία διασπορά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε ακριβώς που βάζουμε τις εξαιρέσεις και οι εξαιρέσεις αυτές ε, να έχουν μια καθολική ισχύ, όχι ε, με άλλα νομοθετήματα να τις ε, ανερούμε αυτές τις εξαιρέσεις είναι, βλέπουμε ας πούμε την εξαίρεση για τα ταμεία σε ένα νομοθέτημα ενώ ε, το RTS δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Επομένως, ε, από τη στιγμή που το RTS και η κατεξουσιοδότηση πράξης δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτές, ε, τότε θα πρέπει να προβλέψει κανείς μία αναφορά για την ημέρα κατά την οποία ή για την θέση σε ισχύ, μετά από την οποία θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει η εξαίρεση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή, πολλά σημαντικά πράγματα αντιμετωπίζει, ούτως ή άλλως ε, είναι γεγονός ότι και εμείς ε, ε, προχωράμε σιγά σιγά γιατί προχωράμε σε έδαφος το οποίο δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ε, απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και πώς έχει όλο το σύνολο του πολιτικού διαλόγου για την κάθε απόφαση. Ε, έχουμε και τους τριγωνικούς διαλόγους. Ε, θα πρέπει το level 1 να γίνει level 2 και αυτό να το κάνουμε με πιο εντατικό ρυθμό. Έχουμε επίσης ε, ε, βάλει ας πούμε στο MIFID ε, την ανάπτυξη, την των μικρομεσαίων εταιριών. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε κάποιους τρόπους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις, την κερδοσκοπία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε ό,τι καταφέραμε και πετύχαμε στο level 1 να μην αναιρεθεί τελικά στο ε, level 2. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα, χρειαζόμαστε τυποποιημένα ε, στοιχεία έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και οι global regulators περί τίνος ε, πρόκειται. γιατί όλα συμβαίνουν πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, ούτε σε τοπική ούτε σε περιφερειακή. Έχω εδώ μία έκθεση σχετικά με την συλλογή δεδομένων το, το FSP και ε, ε, καταλαβαίνουμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ένα σωρό ένα σωρό trade reports τα οποία στην ουσία αναφέρονται σε παρόμοια πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε μία κεντρική έκθεση που να ε, αναφέρει όλα τα στοιχεία αυτά. Τέλος, ε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι μελλοντικές προβλέψεις για τις συντάξεις ε, θα εξαρτηθούν και από τον ιδιωτικό τομέα και όχι πλέον από τον δημόσιο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει με τρόπο ώστε να έχει υψηλότερη επιστροφή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε το μήνυμα αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουμε και την νομοθεσία μας κινούμενη από την πλευρά ας πούμε της προστασίας των ε, καταναλωτών. Ε, δεν θέλουμε να είμαστε απλώς διαφανείς, ε, θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε τους προβληματισμούς και να καλύψουμε τα συμφέροντα του τελικού χρήστη. Όλα αυτά είναι πολλά και προβληματικά σημεία τα οποία αφορούν τα προϊόντα τα επενδυτικά. Ευχαριστώ. Η Άλτε δεν είναι παρούσα. Προχωράμε λοιπόν στην ΚΟΕ. Φάβιο Ντεμάζη, παρακαλώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω ε, στο όνομα της Άλτε, αλλά προσβλέπω στη συνεργασία με όλους σας πάνω στο δύσκολο αυτό θέμα. αυτή τη στιγμή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούμε ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση βλέπουμε να καταραίει ο δανεισμός και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τις κεφαλαγορές. Εγώ θα πρότεινα να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι που η Ευρώπη έχει τραπεζοκεντρικό σύστημα, διότι υπάρχει, οι επιχειρήσει έχουν διαφορετικό μέγεθος, ε, υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, γλώσσε, ιδιαιτερότητε τοπικέ. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούν να κάνουν οι κεφαλαιοχερές όσον αφορά τη χρηματοδότηση μεγάλων εγχειρημάτων, αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε μαγική ράβδο για να ε, λύσουμε το πρόβλημα των επενδύσεων. Εμένα η βασική μου ανησυχία είναι ότι όταν μιλάμε για την Ένωση Κεφάλαια Αγορών δεν μπορούμε να μη μιλάμε για την αγορά ομολόγων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ξενεξετάσουμε θέματα όπως είναι τα ευρωομόλογα με όλες τις νομικές συνέπειες. Δεύτερον, ανησυχώ κάπως για τις διαφωνίες που υπάρχουν όσον αφορά την τυκλοποίηση, διότι ή δεν υπάρχει πρόβλημα με ε, αυτά τα, με αυτούς τους ε, τίτλους, με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, οπότε δεν αρκεί απλά η ζήτηση ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα, για παράδειγμα, του ε, Καναδά, όπου απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται οι ε, τίτλοι, να επανεισάγονται ως ε, ασφάλεια. Μπορούμε να φροντίσουμε να επιμερίζουμε περισσότερο τον κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε τους συστημικούς κινδύνους. Τέλος. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να συζητήσουμε το χρηματοπιστωτικό κταίο και αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε μια τέτοια ιδέα, διότι έχουμε δει στο παρελθόν ότι είναι πολύ ωραίο να έχουμε χρηματοπιστωτικές αγορές ε, που να στηρίζουν τις επενδύσεις, αλλά όταν αναπτύσσονται σε τομείς που δεν συνδέονται με την πραγματική οικονομία μπορεί να εμποδίζουν την ανάπτυξη. Ε, θα χωρώ πολύ να συζητήσω περαιτέρω τα θέματα αυτά μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ Φάμπιο. Σβεν Κίκολτ, ε, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη ακρόαση και προσβλέπω στη συνέχεια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε το ρόλο μας πάρα πολύ σοβαρά. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στείλει ένα μήνυμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για αυτό το θέμα θα είναι κάτι συμβολικό. Γι' αυτό θα ήθελα να συντονιστούμε και με τις συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σύντομα θα υπάρχουν παρόμοιες συζητήσεις και θα είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε το θέμα από κοινού. Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Σκιώδης των Σοσιαλιστών, ότι δηλαδή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κοιτάμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα μόνο μακροπρόθεσμα. Πρέπει να συζητούμε ε, με τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, άλλοι θα είναι ευχαριστημένοι, άλλοι δεν θα είναι κλπ. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι μία πτυχή, σημαντική. Υπάρχει όμως και μακροοικονομική προπτική. Και αυτή η μακροοικονομική προπτική ποια είναι. είναι ποια είναι η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γιατί το έχουμε έχει βοηθήσει να εξυπηρετήσει την πραγματική οικονομία το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχει γίνει αυτό και αυτό ρωτάνε οι πολίτες, αυτό θέλουν να ξέρουν. Θέλουν να ξέρουν είναι τώρα πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να πάρει κανείς δάνειο. Μπορώ να επωφεληθώ από τα κέρδη της τραπεζάς μου, από τις δικές μου επενδύσεις ή όχι ή μήπως το μεγαλύτερο κομμάτι το τρώει η μηπω το μεγαλυτερο κομματι το τρωει η δικαιση η όλων αυτών. Και εγώ παίρνω ψίχουλα. Και είναι βέβαια και το θέμα της χρηματοπιστωτική σταθερότητας και οι πιθανότητες νέας οικονομικής κρίσης. Τέλος, όλο το θέμα της αξιοπιστίας είναι τώρα πιο πιθανό και το βλέπουν έτσι οι αγορές ότι αν πάρει κανείς ένα ομόλογο στην τράπεζα θα λογοδοτήσεις αν πτωχεύσει η τράπεζα. Δηλαδή και εσύ θεωρείς υπεύθυνο ή όχι. Είναι θέμα περιορισμένης εξασφάλισης. Αν πάρω δηλαδή ένα τέτοιο μόλογο περιορισμένης εξασφάλισης, μετά θα είμαι και εγώ υπεύθυνο αν δεν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Υπάρχουν διαφορετικές ιδέες λοιπόν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί κανείς. Δεν θα ήταν καλό να αρκεστούμε σε μία μόνο μελέτη βάσει μιας περίπτωσης. Θυμάμαι πολύ καλά παλιά τα, τις νεοκλασικές θεωρίες και τις μετακεσιανιές και εγώ ήμουνα στη δεύτερη περίπτωση βάσει αυτών ε, σπούδασα γι' αυτό και εξεπλάγει λιγότερο για την κρίση αλλά υπάρχουν διαφορετικές βασικές θεωρίες Συνεπώς πιστεύω ότι όταν κοιτάμε τις μακροοικονομικές προοπτικές δεν πρέπει να αναθέσουμε μία μόνο μελέτη πρέπει να πάρουμε μια απόφαση Πού θα βασιστούμε, σε ποιες περιπτώσεις θα βασιστούμε. Αν λοιπόν πάρουμε μία μελέτη θα βασιστούμε σε μία μόνο περίπτωση και θα ήταν λάθος. Εξάλλου και το κοινό θα έπρεπε να ξέρει ότι ανάλογα με την υπόθεση εργασίας καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα και να ξέρουμε κατά πόσο αυτά συγκλίνουν ή όχι. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα από κάτω προς τα πάνω. Και εδώ είναι που έρχομαι στην αναλογικότητα. Γιατί είναι σαφές. Ακούω συνέχεια τις διαμαρτυρίες, αλλά πρέπει να ξέρουμε τελικά τι είναι αυτό που φέρει σε κίνδυνο τους μικρούς παίκτες. Και τι είναι αυτό που τους επιβαρύνει περισσότερο. Σε όλους τους νόμους υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Αλλά όταν έρθουμε στα άρθρα και στις διατάξεις, εκεί δεν έχει πολλές επιλογές ο επόπτης να δράσει, γιατί τελικά υπάρχει ένας νόμος για όλες τις επιχειρήσεις και δεν αλλάζει τίποτα από το αν έχεις μια ωραία αναλογικότητα στα λόγια, αλλά δεν υπάρχει διαφοροποίηση τα βασικά κείμενα του νόμου. Γι' αυτό χρειάζεται μια ανάλυση από τις επιχειρήσεις αφενός και από την άλλη μεριά μια νομική ανάλυση ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφοροποίηση από τον νόμο και άρα ο φόρτος στους πιο μικρούς παίκτες να μην είναι υπερβολικός. Τέλος, θα ήθελα να δούμε και το τραπεζικό έργο, την ε, σχετική μελέτη που έχει γίνει στη Βουλή των Λόρδων, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Α θυμηθούμε τι συζητήσαμε. Φτάσαμε στο bonus cap. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν για μια άλλη λύση που εγώ προσωπικά βρίσκω ότι έχει πλέον εκτήματα δεν ρυθμίζουν ένα ανώτατο όριο. Αν όμως έχει πρόβλημα η επιχείρηση, τότε ευθύνεται και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για τους μετόχους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και να σκέφτονται το μέλλον στην κάθε τους δράση. Καλό θα ήταν λοιπόν να το δούμε. Τα κίνητρα δηλαδή στην διαχείριση. Συνεπώς λέω στον εισηγητή ότι θα ήθελα οι σκιώδεις με την γραμματεία να συζητήσουμε σε βάθος τι μελέτες χρειαζόμαστε και πώς θα τις ετοιμάσουμε καλά. Επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες να μπουν στη συζήτηση. Ο τίτλος αυτός είναι τόσο μεγάλος που υπάρχει κίνδυνος να το ξεπετάξουμε στα βιαστικά και να χάσουμε την αξιοπιστία που θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο θέμα. Ευχαριστώ. Δεν ήταν πάρα πολύ σύντομη αυτή η παρέμβαση, αλλά έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα. Μόνο ένας ε, σκιώδης και μετά ο εισηγητής μας, ο Μάρκο Τσάνι από το EFTD πρώτα. Ε, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί οι προηγούμενοι συνάδελφοι ήδη ε, ανέφεραν τα πιο σημαντικά ζητήματα και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και πιστεύω ότι το κλίμα είναι θετικό και θα έχουμε πολύ επικοδομητικές ε, συζητήσεις τους επόμενους ε, μήνες μεταξύ μας. Ε, ο εισηγητής και οι εκπρόσωποι διαφόρων πολιτικών ομάδων. Το θέμα είναι σημαντικό και επομένως πρέπει να ε, ε, είμαστε και φιλόδοξοι. Άλλωστε το διακύπαυμα είναι μεγάλο. Και επομένως αυτή η έκθεση θα είναι καλή εάν έχουμε ξεκαθαρισμένα στο μυαλό μας, ξεκαθαρισμένο συγγνώμη στο μυαλό μας, ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι μας, πού στοχεύουμε δηλαδή. Σήμερα το πρωί ε, ακούσαμε και κάποια θέματα όσον αφορά το τι έχει γίνει μέχρι τώρα ε, για την ρύθμιση των κεφαλαίων ε, Ολοκληρώσαμε μία φάση που είναι μία φάση άμεσης δράσης έτσι ώστε ε, να ε, αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις μιας κρίσης. Επομένως, ε, οι αποφάσεις μέχρι τώρα αποφασίστηκαν και ελήφθησαν και υλοποιήθηκαν έτσι ώστε ε, να εξισορροπηθεί μια κρίση. Τώρα όμως ε, θα πρέπει με, το, με, την, ε, με τους κανόνες τους οποίους θα καταρτήσουμε θα πρέπει να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος και θα πρέπει πλέον οι χρηματαγορές να μπουν στην υπηρεσία του γενικού οικονομικού συμφέροντος όσον αφορά ε, την Capital Markets Union. Προφανώς πρόκειται για ένα βήμα θετικό, αλλά προσοχή και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Γκίγκολντ από τους πράσινους ε, ξεκινώντας από την έκθεση αυτή θα πρέπει ε, να αναρωτηθούμε πρώτον, σε τι χρησιμεύει το χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα και δεύτερον, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύω ότι ο ρόλος του ε, θα πρέπει να ε, είναι υποστηρικτικός της χρηματικής οικονομίας. Θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Όταν μιλάμε για Capital Markets Union, βεβαίως καλοδεχούμενη είναι η εναρμόνιση των πλατφορμών, ε, ανταλλαγών και επενδύσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καλοδεχούμενο είναι και ένα σημείο επί του οποίου θα πρέπει να εστιάσουμε και την προσοχή μας. Καλοδεχούμενη λοιπόν η εναρμόνιση των ε, διαδικασιών αφαιρεγγιότητας για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, προσοχή, η χρηματοπιστωτική κρίση προκλήθηκε από υπερβολική χρήση ε, των ε, χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών εργαλείων θα πρέπει να ε, κινηθούμε προσεκτικά. Το να τα μεταφέρουμε όλα πλέον από τα χρηματοπιστωτικά ε, στις κεφαλαιαγορές ε, ίσως είναι εξίσου λάθος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές χωρίς όμως να λειτουργήσουμε πλέον ένα σύστημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάνω κάτω καλά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό το σύστημα, επειδή λειτουργεί περίπου καλά στις Ηνωμένε Πολιτείε, να το ε, να το ε, μιμηθούμε εδώ και να το ε, κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό σύστημα είναι διαφορετικό. Ε, έχει αποτελείται κυρίως από πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αντίθεση με το σύστημα των Ηνωμένων ε, Πολιτειών. Το περιβάλλον εκεί είναι διαφορετικό. Επομένως με δυσκολία μπορώ να δω ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στον οικογενειακό καπιταλισμό σε, σε οικογενειακές εταιρείες ε, με όχι πολύ εκλεπτισμένες γνώσεις ε, του καπιταλισμού και της ε, οικονομίας, πώς μπορεί να ταυτιστεί με τα συμφέροντα ας πούμε των θεσμικών επενδυτών και με τα συμφέροντα των μεγάλων επενδυτών γενικά. Επίσης, να βασιστούμε για την ε, χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ε, σε μόνο μεγάλους ή θεσμικούς επενδυτές νομίζω ότι είναι εσφαλμένη στρατηγική. Στην Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή 70% προσωπική αποταμίευση η οποία επενδύεται μέσω και μακροπρόθεσμα ενώ η θεσμική ε, επενδυτές έχουν πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ε, πρέπει να κινητροδοτήσουμε ε, τις πιο μακροχρόνιες, πιο μακρόθωρες επενδύσεις και θα πρέπει βεβαίως να δούμε ένα, με ποιο τρόπο μπορούμε να λειτουργήσει στις νέες, μέσα στα νέα στοιχεία αυτά ένα <clears throat> τραπεζικό σύστημα, το έδειξε άλλωστε και το έδειξαν και οι, οι τελικές τράπεζες, ε, ένα τραπεζικό σύστημα λέω το οποίο βασίζεται περισσότερο στην ε, ε, ατομική αποταμίευση ε, ε, εμείς ε, μονάχα στο, στην περίπτωση του, της Μοντεπάς και της Χένα αναγκαστήκαμε να κάνουμε τραπεζική εξυγίανση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απλώς χρειάστηκαν κάποιες διορθώσεις. Ένα λοιπόν τραπεζικό σύστημα πιο παραδοσιακό, πιο τοπικό, λιγότερο συνδεδεμένο με τα χρηματοπιστωτικά ε, αυτό είναι ένα, ε, ένας από τους στόχους που πρέπει να έχουμε. Ε, κάτι άλλο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους οι ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτό το shadow banking, το σύστημα το οποίο αποτελεί αυτό το ε, shadow banking. Εγώ δεν ήμουν όταν ξεκίνησε η κρίση βουλευτή στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εσεί προσπαθήσατε να ρυθμίσετε αυτό το shadow banking και τώρα με την ε, Capital Markets Union και με το πράσινο, την πράσινη βίβλο ε, του, της Κομισιόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια ακριβώς γραμμή θέλουμε να ακολουθήσουμε όσον αφορά το shadow banking. Τελευταίο ένα κίνδυνος ο οποίος υφίσταται ακόμη στην ε, ε, Capital Markets Union είναι το εξής. Εάν ε, οθήσουμε την προσωπική αποταμίευση αυτή των οικογενειών προς την κεφαλοαγορά, τότε θα αφαιρέσουμε αυτήν την πηγή χρηματοδότησης από τις τράπεζες μέσω και, και μακροπρόθεσμα ε, οι τράπεζες χρηματοδοτούνται, στηρίζονται στην ε, αποταμίευση των ε, οικογενειών. Εάν λοιπόν πάρουμε τα κεφάλαια αυτά από τις τράπεζες, κινδυνεύουμε να αποσταθεροποιήσουμε το σύστημα και ε, θα οδηγήσουμε και τις τράπεζες ε, στις, ε, χονδρικές, στις συναλλαγές χονδρικής που εξορισμού είναι πιο επικίνδυνες και αμφιβόλου αποτελέσματος από ότι η Λιανική. Αυτά ήθελα να σας πω και πραγματικά ανυπομονώ όπως και άλλοι συνάδελφοι να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χόχμαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ζήτησα το λόγο. Ε, είμαι απλά ένα ταπεινό μέλος της Επιτροπής αυτής. Ε, θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μέρος της συζήτησης αυτής. Θα ήθελα να ευχηθώ στον εισηγητή και τους σκιώδεις σε κάθε επιτυχία. Όταν μιλάμε για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μας ενδιαφέρουν όχι μόνο οι παράγοντες, μας ενδιαφέρουν και οι ρυθμιστές, οι αρμόδιες αρχές και οι νομοθέτες. Κατά κάποιο τρόπο όμως εμείς βρισκόμαστε εκτός των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη δημιουργούμε. Και το λέω αυτό διότι μερικές φορές βλέπουμε τομεακά το θέμα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κάποιοι θεωρούν την χρηματοπιστωτική αγορά ε, ξεχωριστή οντότητα από την πραγματική οικονομία. Εγώ όμως δεν μπορώ να φανταστώ την ε, ε, πραγματική οικονομία χωρίς τράπεζες, τιμολόγια κλπ. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ρευστότητα στην Ευρώπη, τεράστια ρευστότητα, αλλά πολύ χαμηλές επενδύσεις. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση εάν δεν εξετάσουμε τι έχουμε κάνει εμείς και τι αποτελεί δική μας ευθύνη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε δυσκολεύσει το, ε, το να δίνονται δάνεια και το να λαμβάνονται δάνεια. Όταν έχουμε περισσότερη σταθερότητα θα πρέπει να δημιουργήσουμε κατόφλια για τη χρηματοδότηση διότι αυτό αποτελεί μέρος της σταθερότητας. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να αναλαμβάνονται και κίνδυνοι. Όπως ανέφεραν και διάφοροι συνάδελφοι, το να αναλαμβάνει, να αναλαμβάνει κανεί κίνδυνο, το να αναλύει τον κίνδυνο και να επιμερίζει τον κίνδυνο αποτελεί μέρο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε του κανόνε που υιοθετήσαμε εμεί. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό μέρος ε, της συζήτησής μας. Μερικές φορές ο κόσμος νομίζει ότι η Ένωση Κεφαλαιογορών ε, θα αποτελέσει λύση για όλα. Δεν ε, νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό. Στις χρηματοπιστωτικές μας αγορές δεσπόζουν οι τράπεζες. Έχουμε ρυθμίσει τις αγορές αυτές μερικές φορές υπερπολικά καλά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν επενδύσεις, ρευστότητα, αγορές να λαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα ορατό, ότι έχουμε πολύ χαμηλές επενδύσεις ε, σε σχέση με την πολύ υψηλή ρευστότητα που έχουμε. Αυτή η πολύ υψηλή ρευστότητα με τα χαμηλά επιτόκια μπαίνει σε άλλους τομείς της ε, αγοράς αυξάνοντας τις τιμές και το φθηνό χρήμα σε συνδυασμό με τις ε, υψηλές τιμές ε, δημιουργούν φούσκια. Έχουμε λοιπόν τη ζήτηση, δεν έχουμε όμως την προσφορά. Ίσως να είναι πολύ καλή η μετακέινσιανή προσέγγιση όπως υπόθηκε, αλλά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και άλλες οικονομικές σχολές όπως είναι η Αυστρική ή ακόμα και την πραγματικότητα και να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε τις, ε, το πολύ χαμηλό επίπεδο επενδύσεων ε, παρότι έχουμε τόσο υψηλή ρευστότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνιο Ταγιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι στην έκθεση πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου θα πρέπει να φέρεται η τροχιά που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την ε, ε, οικονομία αυτού του είδου. Ε, νομίζω διαφάνει καθαρά και από τη σημερινή συζήτηση. Αυτό που θέλουμε είναι ότι θέλουμε να μα βοηθήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα έτσι ώστε να βοηθήσει μάλλον την πραγματική οικονομία η οποία θα πρέπει να προσπαθήσει να βγει από την κρίση. Ε, δύο πράγματα όσον αφορά τον κανονισμό. Θα πρέπει να αναλύσουμε τη, την επίπτωση ε, της better regulation. Είναι γεγονός ότι έχουν υπάρξει κάποιες επικαλύψεις, κάποια επιπλέον ε, διοικητικά βάρη και κόστη, τα οποία θα πρέπει να σταματήσουν. Θα πρέπει να προβλέψουμε επίσης εάν η Κομισιόν και οι αρχές επιτήρησης έχουν την απαραίτητη ε, πολιτική δικαιοδοσία. Όσον αφορά το άλλο σκέλος, ένας από τους στόχους που πρέπει να έχουμε είναι να συνδυάσουμε το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό με την Τραπεζική Ένωση από τη μία και με το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker από την άλλη. Ε, αναφέρομαι ας πούμε εδώ στο θέμα της χρήσης των συνταξιωτικών ταμείων για τη δημιουργία ε, υποδομών. Νομίζω ότι στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ήδη έχει ε, ε, ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, ο ρόλος των τραπεζών, κυρίως τις λαϊκές τράπεζες, τις συνεταιριστικές τράπεζες που είναι πολύ κοντύτερα στους επενδυτές και στο, συγγνώμη, στον απλό κόσμο και στις μικρές επιχειρήσεις. Η κεφάλαια αγορά βεβαίως είναι σημαντική Απ' την άλλη μεριά και οι τράπεζες είναι εξίσου σημαντικές. Ενδεχομένως θα πρέπει να αναπτυχθούν τα venture capitals. Ε, ωστόσο, ήδη από τώρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη δέσμη COSME, η οποία για πρώτη φορά ε, ε, χρησιμοποιεί τα venture capitals έτσι ώστε να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι και σε άλλες χώρες όπως και στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ έχουμε δει με παρόμοιες ε, συνέργειες πολύ καλά αποτελέσματα. Τελευταίο, ε, η χρήση της κεφαλαιογοράς θα πρέπει να είναι χρήσιμη κυρίως για την πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο ε, για την επίλυση των προβλημάτων πίστης που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει καλά να ελέγξουμε την χρήση του SME Supporting Factor στα πλαίσια της Βασιλείας 3, γιατί το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία, σε συνεργασία και συμφωνία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μπαρνιέ, στον, τον οποίο είχα και εγώ ίδιος ε, στηρίξει, που ε, είχαν δώσει όθηση στις μικρές ε, εταιρείε, στι μικρές επιχειρήσεις ε, που ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλύπτονται στα πλαίσια της Βασιλεία 3 όσον αφορά τέτοιου είδου ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή είναι, πρέπει να είναι μια σταθερή επιλογή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Now for final remarks, the Ο εισηγητής εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και συναδέλφους για την, ε, τις συνεισφορές τους, για τα θέματα τα οποία ανέφεραν. Όλα αυτά τα οποία λέχτηκαν βρίσκουν υποστήριξη σε μένα. Πράγματι, θα πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές σε όλες τις σκέψεις που θα διατυπώσουμε στην έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει επίσης να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την προστασία των καταναλωτών γιατί αυτό είναι τμήμα του καθήκοντος μας ως εκπροσώπων σε μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία. Αυτό μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε η Κέιτ Σουίμπτον ότι πρέπει να υπάρξει συνεκτικότητα μεταξύ του επίπεδου 1 και του επίπεδου 2. Θα πρέπει να διατηρηθεί η συνεκτικότητα που υπάρχει και φυσικά να βελτιωθεί. Και ερχόμαστε εδώ σε ένα κέριο θέμα για μας που θα μας απασχολήσει στους ε, επερχόμενους μήνες. Το θέμα το οποίο έθεσε πίσω ο Σφεν Γίγκολτ Πρέπει να ζητήσουμε μία μελέτη από την Κομισιόν ή πρέπει... Και η Κομισιόν βέβαια μπορεί να διατυπώσει περισσότερες εκθέσεις, αλλά μήπως θα έπρεπε εμείς να ζητήσουμε χωριστές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα και επίσης πώς μπορούμε στην νομοθεσία να εδραιώσουμε μια καλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ μεγάλων και <clears throat> μικρών ε, δανειοληπτών, αυτό είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ιδιαίτερα θετικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Τσάνη προηγουμένως. Η έκθεσή μας έχει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα θεμάτων και γι' αυτό θα είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε φιλόδοξοι. Βλέπω λοιπόν το ρόλο μου ως εισηγητή, ως ένα ρόλο φιλόδοξο. Χαίρομαι που οι σκιώδεις εισηγητές είναι έτοιμοι να συμβάλλουν και επομένως προσβλέπω σε ευρύες συζητήσεις τους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την εξέταση στις 3 Σεπτεμβρίου του σχεδίου έκθεσης και μετά θα έχουμε μια προθεσμία για τροπολογίες και το επόμενο βήμα θα εξαρτάται από τις ε, συζητήσεις μεταξύ του εισηγητού και των σκιωδών. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί στις 6.30 θα ψηφίσουμε την Εύση μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών.